Iniziamo. Innanzitutto. Αρχίζουμε. Καταρχήν. Καλή χρονιά σε όλους. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας σε μια πολύ σημαντική στιγμή και ευκαιρία που μας επιτρέπει να γνωρίσουμε και να αξιολογήσουμε τις θέσεις ε, του Ντάτσαν Τσόλος, του Επιτρόπου που έχει διοριστεί για την ε, γεωργία και την ε, ανάπτυξη της υπέθρου. Σας ευχαριστώ κύριε Τσόλος για την παρουσία σας και σας ευχαριστώ και για τη διαθεσιμότητά σας να απαντήσετε στις ερωτήσεις της ακρόασης. Θέλω όμως να σας πω μερικά πράγματα εισαγωγικά. Η Επιτροπή μας εξέφρασε τις ανησυχίες της για τις κατευθύνσεις του εγγράφου της Κομισιόν για την μεταρρυθμισμένη ατζέντα ε, της ε, συνολικής μεταρρύθμισης και το είχαμε αναφέρει αυτό στην κυρία Φίσερ Μπόλς, την προκάτοχό σα λόγω της περικοπής των κονδυλίων που βλέπαμε εμεί σε αυτό το έγγραφο και ζητήσαμε εμεί η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ να πάρει μια πρωταρχική θέση πολιτικού προβληματισμού. Αλλά αντί γι' αυτό βλέπουμε να έχουμε εδώ έναν ανταγωνισμό πόρων και κονδυλίων που υποβαθμίζει τη Γεωργία και το ρόλο της ε, έναντι των νέων προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει η Ένωση. Τότε μας είχε πει η Επίτροπος ότι το όραμά της δεν ήταν αυτό και ελπίζω και εσείς να επαναλάβετε το ίδιο πράγμα. Επίσης αυτή η Επιτροπή από τη στιγμή που ανέλαβε μπόρεσε να εξετάσει της κρίσης που πλήττουν τους διάφορους γεργικούς τομείς της Ευρώπης τον γαλακτοκομικό τομέα, ο οποίος επλήγει σημαντικά από την αλματώδη μείωση των, σημών, των τιμών. Και βλέπουμε ότι αυτή η κρίση πλήττει όλους τους γεωργικούς τομείς στην Ευρώπη, από το βορρά στο νότο, από την Ανατολή στη Δύση. Θεωρούμε λοιπόν ότι εμείς μπορούμε να αναπτύξουμε μία γεωργία σύμβατη με τις ανάγκες της ευρωπαϊκής κοινωνίας, σεβόμενη τις ανάγκες των πολιτών και των γεωργών των οικονομικών 27 κρατών μελών. Θέλω τώρα να σας αναφέρω τα διαδικαστικά αυτής της ακρόασης. Να σας ε, θυμίσω ότι βάσει των προσανατολισμών για την εκλογή της Κομισιόν, παράρτημα 17 του κανονισμού, το Κοινοβούλιο κρίνει τους επιτρόπους βάσει του ευρωπαϊσμού τους, ε, της ανεξαρτησίας και τις ε, γνώσεις του χαρτοφυλακίου τους, όπως επίσης και την ικανότητα επικοινωνίας. Θέλω να σας θυμίσω ότι πριν από την ακρόαση, ο υποψήφιος επίτροπος απάντησε γραπτός σε ένα αρχικό ερωτηματολόγιο το οποίο έχει δοθεί ήδη στους βουλευτές σε όλες τις γλώσσες. Λοιπόν, Κατά πρώτον, ο υποψήφιος επίτροπος θα κάνει μία εισαγωγή που δεν θα ξεπεράσει τα 10 λεπτά. Θα ακολουθήσουν μετά 2 ώρες και 40 λεπτά ερωτήσεων με έναν πρώτο κύκλο τοποθετήσεων ενός εκπροσώπου για κάθε πολιτική ομάδα. Η συζήτηση θα γίνει σύμφωνα με το σύστημα ping-pong για πέντε λεπτά η κάθε φάση. Ένα λεπτό για, για κάθε ερώτηση, δύο λεπτά για την απάντηση του Επιτρόπου, ένα λεπτό για ανταπάντηση αν χρειαστεί φυσικά και ένα λεπτό για την τελική απάντηση, αν πάλι χρειαστεί. Ο χρόνος των βουλευτών είναι ένα λεπτό. Πιο σύντομες θα είναι οι ερωτήσεις, περισσότερο χρόνο θα έχουμε στη διάθεσή μας για να απαντήσει ο υποψήφιος επίτροπος και για να ακολουθήσουν και άλλες ερωτήσεις. Οι απαντήσεις θα πρέπει να, συγγνώμη, οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι μέσα στο θέμα των αρμοδιοτήτων του επιτρόπου και δεν θα πρέπει να επευκεύουν σε άλλα αντικείμενα. Η συζήτηση θα έχει διερμηνία σε 22 γλώσσες. Όλοι οι ομιλητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη μητρική τους γλώσσα. Η συζήτηση μέσω του web stream αναμεταδίδεται απευθείας ε, στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Επίσης, θα έχουμε ένα πλήρες πρακτικό το οποίο θα το έχετε στη διάθεσή σας το συντομότερο. Λοιπόν τώρα αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε θέλω να δώσω το λόγο στον Τάτσαν Τσόλος ε, για να μιλήσει για 10 λεπτά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε με κύριε Πρόεδρε Τεκάστρο, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, κυρίε και κύριοι. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι εδώ σήμερα το πρωί. Γιατί με την έναρξη ισχύω τη συνθήκη τη Λισαβόνα, η οικογένεια των ε, υπευθύνων για την ανάληψη αποφάσεων ε, έχει ενισχυθεί. Είστε επίσης υπεύθυνοι για τις αποφάσει που λαμβάνονται σε αυτή την πολιτική πλέον και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αν με επικυρώσετε θα ακολουθήσω αυτή τη στρατηγική λαμβάνοντα υπόψη τη νέα αυτή πραγματικότητα. Και γιατί με ικανοποιεί αυτό, διότι γνωρίζω ότι η ποιότητα και η Τη κοινή γεωργική πολιτική θα ενισχυθεί με τη δική σα συμβολή και με την ε, στεναρή σα συνεργασία. Γνωρίζω ορισμένου από εσά από τι προηγούμενε μου ε, ευθύνε ω Υπουργού ε, Γεωργίας της Ρουμανίας ή από άλλε ευκαιρίε κατά τη διάρκεια τη επαγγελματική μου ζωή. Γνωρίζω πω η ποικιλομορφία τη Ευρωπαϊκή της Ευρωπαϊκής και των περιοχών τη Υπέθρου αντιπροσωπεύεται εξαίρετα εδώ. <clears throat> Η Επιτροπή αυτή αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα πολυμορφίας διαφοροποίησης που θέλω να διατηρήσω και να προωθήσω στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Επίση πιστεύω πως αυτή ε, η Επιτροπή αποτελεί έναν πολύτιμο πόρο για την γεωργία και για τις γεωργικές πολιτικές. Ως πολιτικός είμαι ανοιχτό στις απόψεις και τις ιδέες σας και από αυτό το πνεύμα θα ήθελα να με αξιολογήσετε και να έχουμε έτσι και μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, ώστε να σας παρουσιάσω τις ιδέες μου και να έχουμε και μια πρώτη αίσθηση για το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ε, είμαι έτοιμος να σας ακούσω και να σας δώσω τις ιδέες μου, αλλά πριν από αυτό παρακαλώ να με επιτρέψετε να σας ε, ε, συστηθώ και να σας παρουσιάσω κάποιες από τις ιδέες όσον αφορά το μέλλον της εντολής μου και επιτρέψτε μου να το πράξω στη γλώσσα μου στα ρουμανικά. Εγώ γεννήθηκα το 1969 στην Ρουμανία, μια χώρα που γνώρισε την κολεκτιβοποίηση και την εθνικοποίηση και που πλέον σήμερα έχει βρει τη θέση της στην Ευρώπη. Εγώ ξεκίνησα την καριέρα μου μετά το 1990 και υπό το άστρο της προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εισόδου της χώρας μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υπεπιθύσεις μου είναι άμεσα προσδεδεμένες με τις θεμελιώδεις αξίες της ελευθερίας αλλά και του ενδιαφέροντός μου για την γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Είναι θέματα τα οποία εγώ έχω ε, γνωρίσει εργαζόμενος στον τομέα της γεωργίας είτε εργαζόμενος στις ε, ε, οικογενειακές γέες είτε συνεργαζόμενος με αγροτικούς συνεταιρισμούς και γεωργικά συνδικάτα. Εγώ εργαζόμενος στον τομέα της γεωργίας πάντοτε απαιτούσα ε, να ε, πληρούνε όλοι τις απαιτήσει και πάντοτε έβγαινα από το γραφείο μου. Πιστεύω ότι η γεωργία δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται αντιληπτό από ένα γραφείο, χρειάζεται επαφή επιτόπου. Σύμφωνα με τη συνθήκη της ε, Ρώμης η ΚΑΠ πρέπει να εξασφαλίζει την αυτάρκεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα αξιοπρεπές εισόδημα για τους παραγωγούς. Η ΚΑΠ πάντοτε προσαρμόστηκε στις εσωτερικές και στις διεθνείς προκλήσεις και εξελίξεις. Αλλά παρόλα αυτά τίποτα από τα κεκτημένα που έχουμε σήμερα είναι κάτι το δεδομένο. Η αυτάρκεια δεν είναι δεδομένη σήμερα. Η Ευρώπη έχει σήμερα 27 μέλη, έχει κερδίσει σε διαφορετικότητα και στον τομέα της γεωργίας και στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Η γεωργία δεν είναι μόνο παραγωγός τροφίμων, είναι παραγωγός αγαθών για την πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Γιωργός συμβάλλει όχι μόνο στην διατροφή, συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. συμβάλλει στην προστασία του κλίματος. Γι' αυτό λοιπόν εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει ένας από τους στόχους της, τωρινής, της νέας επιτροπής μάλλον είναι να ορίσει τους στόχους μετά το 2013. Οι Ευρωπαίοι γεωργοί απαιτούν σταθερότητα και οι καταναλωτές θέλουν ασφαλή τρόφιμα. Ο φορολογούμενος θέλει να έχει τη σιγουριά ότι το χρήμα του ξοδεύεται αποτελεσματικά και με διαφάνεια. Θα πρέπει λοιπόν η ΚΑΠ να έχει και την απαραίτητη πρικοδότηση που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας. Η μελλοντική ΚΑΠ θα πρέπει να παραμείνει μια δίκαιη ευρωπαϊκή πολιτική που θα βασίζεται σε τρία στοιχεία. Καταρχήν, οι άμεσες πληρωμές οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για τη σταθερότητα του εισοδήματος των γεωργών. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Φυσικά θα πρέπει να αναλύσουμε με ποιον τρόπο θα καταμνέμονται οι άμεσες επιδοτήσεις με νέες ρεαλιστικές βάσεις. Χρειαζόμαστε μία σύγκληση και μία ισοτιμία μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών γεωργών των διαφόρων περιοχών των κρατών μελών και κρατών των μελών. Νέα οργάνωση των μηχανισμών των αγορών που θα πρέπει να προσεγγίσουν τους στόχους της ΚΑΠ. Πρέπει να διορθώσουμε τις τρευλώσεις της αγοράς και να ανταποκριθούμε τάχιστα και ευέλικτα σε αυτά τα σκαμπανεβάσματα των τιμών που επηρεάζουν και τα εισοδήματα των γεωργών αλλά και το πορτοφόλι των καταναλωτών. Θα πρέπει λοιπόν η αγορά να παίζει ρυθμιστικό ρόλο, αλλά δεν θα πρέπει να έχουμε διακοιμάνσεις οι οποίες θα αποστεθαροποιούν την Ευρωπαϊκή Γεωργία και τα εισοδήματα των Γεωργών. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι μία λύση για το μέλλον η επανάληψη της χρήσης των παλιών μηχανισμών της αγοράς. Διότι βλέπουμε ότι η κατάσταση έχει αλλάξει. Έχουμε κερδοσκοπικά κεφάλαια, νέα κερδοσκοπικά κεφάλαια στην αγορά. Έχουμε τις, ε, ε τις νέες χώρες που αναδύονται και κατακλείζουν την αγορά με νέα προϊόντα. Πρέπει να δούμε την ανάπτυξη της υπαίθρου η οποία θα πρέπει να συμβάλλει στην αναδιάρθρωση και τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις κλιματικές αλλαγές και να στοχεύει στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος. Θα πρέπει να εξέρει τη διαφορετικότητα και την ιδιαιτερότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας να αναπτύξει την τοπική διανομή, την τοπική διαφορετικότητα. Και αυτό με έναν τρόπο πιο έντονο και πιο ορατό. Λοιπόν, ποιότητα και διαφορετικότητα και αυτό θα είναι το πλεονέκτημά μας στις διεθνές αγοράς. Θα πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί στις διαπραγματεύσεις με αυτό το επιχείρημα στο χέρι μας. Ποιότητα λοιπόν και ιδιαιτερότητα των γεωργικών προϊόντων της Ευρώπης και αυτό θα το παλέψω σε συνεργασία με τους συναδέλφους μου και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν μιλάμε εμεί για την ΚΑΠ δεν μιλάμε μόνο για το φαγητό μας, για την τροφή μας. Αλλά μιλάμε και για εκατομμύρια θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θα πρέπει να συνεργαστούμε για να θέσουμε τις βάσεις της Ευρωπαϊκής Γεωργίας του αύριο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που σεβαστήκατε το χρόνο σας και σας ευχαριστώ και για, τις, ε, την αρχική σας ε, τοποθέτηση. Λοιπόν, οι συντονιστές των ομάδων. Ο Άλμπερτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος του, της ομάδας του ΕΛΚ θα ήθελε να καλωσορίσω τον υποψήφιο Επίτροπο και να του ευχηθώ κάθε επιτυχία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Σε σχέση με τους ε, πολλούς τομείς και τις δύσκολες ε, καταστάσεις που επικρατούν, πώς σκοπεύετε να διασφαλίσετε το εισόδημα για τον αγροτικό πληθυσμό της Ευρώπης. Και σημαντικό ρόλο επίσης θα είναι το άρθρο 70 είναι το άρθρο 70 και 72 του κανονισμού 73. Είσαστε κατά της ε, αποχώρηση από το δεύτερο πελώνα κάποιων περιφερειών. Πώς θα τοποθετηθείτε έναντι στις μικρόμεσαίες επιχειρήσεις και καθοριστικό ερώτημα, πώς θα αφήσετε το Κοινοβούλιο να συμμετάσχει στην ε, διαδικασία αυτή προκειμένου να μπορέσει να ασκήσει και την υποπτική του ενέργεια και ε, αρμοδιότητα ο Επίτροπος. Πιστεύω ότι η απάντησή μου στο ερωτηματολόγιο σας ήταν σαφής. Και η τοποθέτησή μου νομίζω εξέφρασε σαφώς το γεγονός ότι η ΚΑΠ θα πρέπει να διασφαλίζει πρώτα απ' όλα το εισόδημα των αγροτών για να διασφαλίζει δηλαδή και τη σταθερότητα της γεωργικής παραγωγής. Εγώ σας το είπα ότι ο πρώτος πυλώνας και οι άμεσες πληρωμές θα πρέπει να διασφαλίζουν τη σταθερότητα του γεωργικού εισοδήματος και θέλω να συνεχίσω προς αυτήν την κατεύθυνση. Τώρα για τα μέτρα ρύθμισης της αγοράς που έχω κατά νου χωρίς να έρχομαι σε μηχανισμούς του παρελθόντος. Αυτοί λοιπόν οι μηχανισμοί θα, ε, θα έχουν ως στόχο την αποφυγή των διακυμάνσεων στην αγορά. Για την ανάπτυξη της υπαίθρου τώρα στο δεύτερο πυλώνα, η ανάπτυξη της υπαίθρου θα πρέπει να παραμείνει στον τομέα της γεωργίας. Δεν μπορούμε εμείς να ξεχωρίσουμε την γεωργική ανάπτυξη από την ανάπτυξη της υπαίθρου. Είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένες αυτές οι δύο έννοιες. Φυσικά θα πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου τη συνοχή μεταξύ των δύο, να μην μένει τίποτα ακάλυπτο. Αλλά θα πρέπει να οικοδομήσουμε τον δεύτερο πυλώνα λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την άμεση ανάγκη εξυγχρονισμού της γεωργίας χωρίς να αφήσουμε έλεγα τίποτα ακάλυπτο. Η συνεργασία για μένα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ουσιαστική, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι σε αυτήν την Επιτροπή υπάρχουν άνθρωποι με τεράστιες ικανότητες των οποίων τη βοήθεια εγώ χρειάζομαι. Άλμπερτ, θες να απαντήσεις? Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την ε, απάντησή σας. Αυτό που θα είναι καθοριστικό την επόμενη περίοδο να υπάρχει και σωστή εξωτερική προστασία. Και ξέρουμε ότι μειώνεται η εξωτερική προστασία, αλλά απαιτείται, ε, απαιτούνται πάρα πολλά σε ό,τι αφορά τους Ευρωπαίους αγρότες. Θα ταχθείτε στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου οι εισαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρούν τις ίδιες, ε, τους ίδιους όρους. Δεν είναι δυνατόν να είναι τόσο αυστηροί οι όροι στο εσωτερικό της Ένωσης και να μην τηρούνται στις εισαγωγές και σε ό,τι αφορά το μέλλον της αγροτικής πολιτικής. Είναι σημαντικό αυτό που συμβαίνει και στην Αυστρία και εδώ θα ήθελα λοιπόν μία απάντηση για το πώς σκοπεύετε να αντιδράσετε γιατί υπάρχουν μεγάλα προβλήματα εισοδήματο και θα είναι σημαντικό να βρούμε απαντήσεις προκειμένου να διασφαλιστεί το μέλλον όλων των ανθρώπων. Σας ευχαριστώ. Είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς έχοντας μόνο ένα λεπτό στη διάθεσή του. Η εξωτερική μας προστασία σε σχέση με αυτό που έχει να κάνει με την ασφάλεια των τροφίμων σχετίζεται και με το, τις συμφωνίες με τους εταίρους τους οποίους ε, συνεργαζόμαστε. Οι απαιτήσει ε, για μια ολόκληρη σειρά τομέων ε, ώστε να έχουμε μεγαλύτερη προστασία θα εφαρμοστεί για όλους τους τομείς. Απαιτούμε οι προδιαγραφές που ισχύουν για τους Ευρωπαίους γεωργούς να ισχύσουν και για τους εταίρους μας. Και όσον αφορά τα γαλακτοκομικά προϊόντα, αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό εξέλιξη μια συζήτηση σε σχέση με το μέλλον αυτού του τομέα με στόχο τον εντοπισμό ενός νέου μηχανισμού που θα μας επιτρέψει να εγκαταλείψουμε το σύστημα των ποσοστώσεων και να εισάγουμε νέους μηχανισμούς. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστώ, Άλμπερντε, ε, σας ευχαριστώ, Επίτροπε, και δίνω αμέσως το λόγο στο Λουίς Καπούλας Σάντος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, εξ ονόματο τη Σοσιαλιστική και Δημοκρατική Ομάδα, θα ήθελα να σα καλωσορίσω και να σα ευχηθώ κάθε επιτυχία. Όπω γνωρίζετε, με τη συνθήκη τη Λισαβόνα και με την ολοκλήρωση τη διαδικασία του phasing in των νέων, των νέων κρατών μελών το 2013, έχουμε μια ιστορική ευκαιρία για να καθορίσουμε τον νέο ρόλο τη γεωργική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συμβατότητα με τον ΠΟΕ με ισότιμο τρόπο. Εδώ λοιπόν εντάσσεται και η ερώτηση, η απάντηση που έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την νέα ισορροπία ανάμεσα στι διάφορες κατηγορίε των γεωργών και ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη και έχει υποδείξει την πρώτη αυτή πολιτική προτεραιότητα. Ω τεχνικό που είστε γνωρίζετε καλά τα στοιχεία όπω και εγώ και ξέρετε τι μεγάλε ανισότητε που υπάρχουν και που προκαλούν την άνεση κατανομή των ενισχύσεων. Και ήθελα λοιπόν να μου πείτε αυτή την αντίφαση που υπάρχει ανάμεσα στην απάντηση που δώσατε γραπτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου εκδηλώνεται μια σαφής πολιτική βούληση για μεταρρύθμιση και άλλες δικές σας δηλώσεις που έχουν αναφερθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη και που αντίθετα μόνες γίνεται λόγος για απλές προσαρμογές φαίνεται να εμφανίζεστε ότι φοβάστε ακόμα και να αναφέρετε τη λέξη μεταρρύθμιση. Λοιπόν, ποιο από τα δύο είναι η πραγματική σας άποψη, Επίτροπε, ο Επίτροπος. Κοιτάξτε, δεν ξέρω ακριβώ σε τι αναφέρει ο τύπο πανευρωπαϊκά, αλλά κύριε Καπούλα Σάντο, θα έχουμε πολλέ φορέ ε, την ε, ευκαιρία να το συζητήσουμε, αλλά ναι, ναι, ήμουν και σαφή. Η γεωργική πολιτική σίγουρα θα πρέπει να προσαρμοστεί καλύτερα στο σημερινό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ενώση των 27. Η κατάσταση του γεωργικού τομέα και τη υπαίθρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει. Υπάρχει μεγαλύτερη διαφοροποίηση και ακριβώ από αυτό το πρίσμα τα έσοδα των γεωργών και η διασφάλιση αυτών των εισοδημάτων ε, μέσω των μεταρρυθμίσεων είναι θεμελιώδη σημασία. Κατά την άποψή μου, μεταρρύθμιση δεν σημαίνει μείωση τη οικονομική ενίσχυση ή η εξάλληψη ορισμένων ε, μηχανισμών. Μεταρρύθμιση σημαίνει προσαρμογή ώστε να σταθούμε στο ύψο τη νέα κατάσταση. Ε, και επειδή περί αυτού πρόκειται, σα εγγυώμαι ότι αυτή θα είναι και η πρόθεσή μα. Ότι δηλαδή να γίνουν οι μεταρρυθμίσει για να μπορέσουμε να βρούμε λύσει προσαρμοσμένε στη σημερινή κατάσταση. αυτή η προσέγγιση μου θα αφορά ολόκληρη την γεωργική πολιτική, αλλά και τις διεθνείς ε, πραγματεύσεις όπου η γεωργία αποτελεί βασικό στοιχείο. Δεν μπορούμε να φανταστούμε διεθνή συμφωνία χωρίς να ε, λαμβάνουμε υπόψη τη γεωργία. Προσπαθούμε πάντοτε να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις ώστε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που μας προσφέρει η διεθνής αγορά. Αυτή είναι η δική μου πραγματικότητα κύριε Καπούλα Σάντος. Δεν ξέρω αν σας απάντησα στην ανησυχία σας, αν σας κάλυψα, αλλά μπορώ να σας εγγυηθώ ότι θα συνεχιστεί ο διάλογος με το Ευρωπαϊκό ε, ε, Κοινοβούλιο. Δεν θα γίνει μέσω του τύπου, αλλά πρόσωπο με πρόσωπο διάλογος αυτό. Ε, Λουίς, θες να κάνεις επερώτηση, ναι. Μια ερώτηση που θα ήθελα να διευκρινίσετε καλύτερα το θέμα το πιο λεπτό, το πιο ευαίσθητο στη διαδικασία μεταρρύθμισης της ΚΑΠ που θα γίνει ε, προσεχώς θα είναι το θέμα των κριτηρίων για την κατανομή των ενισχύσεων. Και γι' αυτό το ζήτημα θα ήθελα να μου απαντήσετε με πολύ συγκεκριμένα. Θεωρείτε ότι το ιστορικό κριτήριο είναι πλέον καταδικασμένο ή ότι υπάρχουν όροι για τη συντήρηση, διατήρηση ορισμένων ε, στοιχείων αυτού του κριτηρίου για μετά το 2003. Ποιε θα πρέπει να είναι κατά την άποψή σα, ποια θα πρέπει να είναι τα νέα κριτήρια για την κατανομή των ε, ενισχύσεων. Συμφωνείτε ότι το περιβάλλον και η απασχόληση μπορούν να είναι δύο εναλλακτικέ ή πιστεύετε ότι υπάρχουν και άλλε. Και τέλο, επειδή πολύ επιφανειακά ε, θίξατε το θέμα του ΠΟΕ στην απάντησή σας. Θα ήθελα λακωνικά να μου πείτε ποια είναι τα ζητήματα που για την υπεράσπιση της ε, ΚΑΠ, της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, θεωρείτε ότι δεν μπορείτε να διαπραγματευτείτε. Ο Επίτροπος. Τα κριτήρια για την κατανομή των ενισχύσεων και η μεταρρύθμιση που θα ήθελα να προτείνω θα έχει στόχο να εγγυηθεί και να προωθήσει μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην κατανομή των ε, γεωρικών ενισχύσεων των ε, που απευθύνονται στις περιφέρειες και στα κράτη-μέλη. Η ιστορική αναφορά δεν νομίζω πως θα είναι η κατάλληλη λύση. Αυτή χρησιμοποιήθηκε όταν ε, θέλαμε να υπάρξει ε, ικανοποίηση των, ε, της κατανομής. Αυτή τη στιγμή όμως η λύση αυτή δεν θεωρώ ότι είναι η καταλληλότερη. Θα πρέπει να αναζητήσουμε νέα ισορροπία. Και έτσι θα σκεφτούμε με συνέπεια τα κριτήρια που θα μας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουμε με καλύτερο τρόπο τα κονδύλια που θα έχουμε στη διάθεσή μας ε, και τις ε, ενισχύσεις και επίσης θα μπορέσαμε να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα σε σχέση με τα κριτήρια ε, που αφορούν το περιβάλλον και την απασχόληση. Αυτοί οι δύο παράγοντες είναι πολύ σημαντικοί και όσον αφορά τον ΠΟΕ να σας πω πως η η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει κάνει σημαντικές ε, πρόοδους και περιμένουμε πως και οι εταίροι μας θα τις ε, κάνουν το ίδιο και ε, θα προχωρήσουμε με ένταση, με ένταση και στις διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει τώρα Μάρτιν Όσλινγκ. Μάρτιν. Να σας καλωσορίσω και εξ ονόματος των Πρασίνων, Θα να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία, αλλά θα θέλαμε πιο συγκεκριμένες απαντήσεις στο μέλλον. Πώς θα προωθήσετε τη βιώσιμη γεωργία, τη, τη διάστατη της βιοποικιλότητας, της αλλαγής του κλίματος, πώς θα τα εμπλέξετε στις άμασες πληρωμές. Και επίσης μιλήσατε για την ευρωποιημένη ε, γεωργία και ως υπουργό στην Ρουμανία ταχθήκατε υπέρ των μικρών αγρατών. Σκοπεύετε να διατηρήσετε και να ελέγξετε τη συνισορροπία και στις άμεσες πληρωμές σε ό,τι αφορά το ποσοστό των επιχειρήσεων και το θέμα των θέσεων εργασίας αναφέρεται προηγουμένως και το εκτιμώ αυτό και αυτό θα είναι, κριτό, θα είναι και το κριτήριο για τα μελλοντικές σας εργασίες. Και μια ερώτηση για το θέμα του γάλακτος. Θεωρώ ότι πρέπει να λάβουμε πιο συγκεκριμένες ε, απαντήσεις. Μπορείτε να φανταστείτε συγκεκριμένους μηχανισμούς για να ρυθμιστεί η προσφορά και μετά το 2013 και θεωρείτε ότι η προώθηση, η ενίσχυση των εξαγωγών αποτελεί και αυτό ένα μέτρο, ένα μηχανισμό για την πρόθεση του κλάδου. Ο Επίτροπος θα απαντήσει. Ευχαριστώ για την αλλαγή του κλίματος και σε ό,τι αφορά την ε, βιοπικιλότητα και τις άμεσες ενισχύσεις. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε να συνεχιστεί και αυτή η συμπερίληψη των κριτηρίων αυτών στις άμεσες πληρωμές, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ρυθμιστεί καλύτερα δεύτερος πυλώνας της ΚΑΠ, προκειμένου να συμπεριληφθούν και στην γεωργία μηχανισμοί για την προστασία της αλλαγής του, κατά του αλλαγής του κλίματος και της ε, Δύο ποικιλότητες. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καλύτερα λοιπόν τα μέσα του δεύτερου πυλώνα για την ΚΑΠ. Τώρα, για τους μικροεκμεταλλευτές τόσο κατά την κατανομή των άμεσων πληρωμών, αλλά και σε άλλα θέματα θα πρέπει να επιδιώξουμε αυτή την ισορροπημένη προσέγγιση. Θεωρώ ότι και εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα του δεύτερου πυλώνα και να καταδείξουμε ότι υπό συγκεκριμένου όρου μπορούν να είναι ανταγωνιστικέ αυτέ οι μικρέ επιχειρήσει, οι μικρέ εκμεταλλεύσει, γιατί οι παραγωγέ του μπορούν να προσαρμοστούν στι συγκεκριμένε τοπικέ ανάγκε και νομίζω ότι εδώ υπάρχουν πολλά περιθώρια στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα όπου φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε πρώτη φάση θα πρέπει να είναι ισορροπημένη η ενίσχυση. Θα πρέπει φυσικά να υπάρχουν να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια, αλλά αυτά θα πρέπει να διαμορφωθούν από κοινού. Δεν μπορώ να επισέλθω σε λεπτομέρειες, δεν έχω αποφασίσει ε, οτιδήποτε και δεν μπορώ να δώσω τέτοια εντύπωση. Αλλά φυσικά από κοινού θα διαμορφώσουμε τους αντίστοιχους μηχανισμούς. Για τον τομέα του γάλακτος θα πρέπει να βρούμε μηχανισμούς και τρόπους προκειμένου ο έλεγχος, ο διοικητικός, να μην υπάρχει διοικητικός έλεγχος της ζήτησης, να ρυθμίζεται αυτόνομα στον κλάδο η ζήτηση. Νομίζω ότι η ομάδα για τον, την παραγωγική παραγωγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνει σημαντική δουλειά γιατί μπορεί να καταρτήσει προγράμματα ανά κλάδο και να ρυθμίσει τα πράγματα μεταξύ των φορέων. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μία λύση. Και επίσης είμαι τεθειμένος να συζητήσω και με τους συναδέλφους για τον ανταγωνισμό σε ό,τι αφορά διάφορους μηχανισμούς που θα εγγυηθούν αυτή την ισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς χωρίς να επισέλθουμε όμως σε λεπτομέρειες και σε ρυθμίσεις της ζήτησης όπως το παρελθόν. Ευχαριστώ. Δεύτερη ερώτηση, κύριε Πίτροπε. Ίσως θα μπορούσατε να απαντήσετε σε ό,τι αφορά την, ε, ε, τις ενισχύσεις των εξαγωγών, γιατί είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα αυτό για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής. Η προκάτοχό σας ε, επικεντρώθηκε σε θέματα απελευθέρωσης σε ό,τι αφορά τις παγκόσμιες αγορές. Θα συνεχίσετε την πολιτική αυτή ή θα προβείτε σε κάποιες συγκεκριμένες ε, διορθώσεις. Όπως σε άλλους τομείς, όπως το χρηματοπιστωτικό τομέα, προκειμένου από πλευράς πολιτικής να προκύψουν πιο πολλοί κανόνες, να μην αφήσουμε την ελεύθερη αγορά από μόνη της να ξεφύγει. Αυτό λοιπόν θα ήταν σημαντικό να το ακούσουμε. Και ύστερα συναντήθηκαν οι Υπουργοί Γεωργίας πρόσφατα στο Παρίσι και υποστήριξαν την ε, γραμμή αυτή. Πώς το αξιολογείται αυτό το γεγονός δηλαδή ότι δίνεται μεγαλύτερος ρόλος πλέον και στην πολιτική και όχι μόνο στην ελεύθερη αγορά. Απάντησε ο Επιτροπός. Ευχαριστώ. Ναι, σίγουρα. Στον τομέα των τροφίμων η αγορά είναι πολύ σημαντική, όπως και στους άλλους κλάδους άλλωστε, αλλά η γεωργία και ο τομέα των τροφίμων έχει και ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό και νομίζω ότι χρειαζόμαστε μηχανισμούς ε, ρύθμισης της αγοράς που δεν θα αντιταχθούν όμως την αγορά, απλά θα την ενισχύσουν. Άρα, ναι, προς αυτή την κατεύθυνση σκοπεύω να συνεχίσω. Για τις ενισχύσεις τώρα των εξαγωγών δεν ε, θεωρώ ότι αποτελεί ουσιαστική λύση για το μέλλον αυτό σε κάποιους τομείς. Ασφαλώς, ασφαλώς οι ενισχύσεις αυτές ε, θα διατηρηθούν. Και θα δούμε τι θα προκύψει και από τις διεθνείς ε, διαπραγματεύσεις Δισκοπεύω ωστόσο να κινηθώ προς την κατεύθυνση της απελευθέρωσης της αγοράς μόνο και μόνο για την απελευθέρωση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ωραία, Επίτροπε. Τώρα το λόγο έχει ο Τζέιμς Νίκολσον. Τζέιμς, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε, ψήφι Επίτροπε. Όταν εγώ έγινα, μέλο έγινα μέλος αυτής της Επιτροπής πριν από 21 χρόνια, διανύω το 21ο, η ΚΑΠ ήταν πάνω από 50% του προπολογισμού. Αν σήμερα σας συγκρίνουμε και αναλάβετε την θεία σας, πουφ, βλέπετε να έχει φτάσει ο προπολογισμό όταν θα φύγετε πια. Γιατί αν δεν υπάρχουν τα χρήματα στον προπολογισμό δεν μπορούμε να έχουμε ούτε το γεωργό ούτε την ε, γεωργική αγροτική οικονομία. Έπειτα, εχθέ επέβαλα κάποιε ερωτήσει στον κύριο Ντάλη και πρέπει να πω ότι δεν ικανοποιήθηκα με τι απαντήσει στι ερωτήσει που του έδωσα και που οι συνάδελφοι σε αυτήν την επιτροπή του έθεσαν. Εκείνο θα συνεχίσει με την ίδια δρομή τη ε, DG Sanko όσον αφορά τι οδηγίε για το έδαφο, δίνοντα στου γεωργίε ορλάνε και περισσότερη γραφειοκρατία και προβλήματα ε, επί τόπου. Τι θα κάνετε θα υπερασπιστείτε την Επιτροπή Γεωργίας στο σύνολο των Επιτρόπων, απέναντι στο σύνολο των Επιτρόπων. Σήμερα μα παρουσιαστήκατε ω μεταρρυθμιστής και ως ε, ε, συνδεδεμένο με τις άμεσες πληρωμές. Πώς θα διασφαλίσετε ότι η κατανομή, η χρηματοδότηση του ΣΚΑΠ θα δίνεται στους ενεργούς γεωργούς και ποιοι είναι ακριβώ οι ενεργοί γεωργοί. Επίτροπε. σε σχέση με τον προπολογισμό, Πιστεύω πως ήταν πολύ ξεκάθαρο. Έδωσα απαντήσεις ε, γραπτός προς το Κοινοβούλιο. Εγώ πιστεύω πως ο προπολογισμό επιτρέπει την βασική λειτουργία της, κοινής, της, της ΚΑΠ. Είναι πολύ σημαντικό ότι θα να διατηρηθεί αυτός ο προπολογισμό. Ένας προϋπολογισμός ε, συνεπής και συνεκτικός. Μπορώ αυτό να το εγγυηθώ και στο πλαίσιο του Συμβουλίου να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε επιχειρήματα για να δικαιολογήσουμε την ε, ύπαρξη ενός σημαντικού γεωργικού προϋπολογισμού. Θέλουμε να έχουμε μια συνεπή, συνεκτική κάπα που να εγγυάται όχι μόνο την διατήρηση των αγορών αλλά και μια ολόκληρη σειρά άλλων κοινών αγαθών που είναι σημαντικά για του φορολογούμενου, χρειάζεται αυτή η στήριξη οικονομική προ τη Γεωργία. Από αυτή την άποψη είμαι πολύ ξεκάθαρο. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε συνεπή κάπου για το μέλλον, εάν δεν έχουμε τα απαραίτητα κονδύλια που θα μας ε, βοηθήσουν να ανταποκριθούμε σε κάτι τέτοιο. Σε σχέση με τη γραφειοκρατία και συγκεκριμένα μέτρα, ε, σε σχέση με το ρόλο των Γεωργίων, εγώ έκανα ήδη θα, θα, θα πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια, ήδη έχει έχει γίνει προσπάθεια για απλοποίηση της ΚΑΠ, αλλά και θα συνεχιστεί, ιδιαίτερα όσον αφορά τους διάφορους πυλώνες και τους τρόπους απλοποίησης της ε, πολιτικής, ε, χωρίς όμως να αποδυναμωθεί η δυνατότητα ελέγχου και οι διοικητικές δυνατότητες. Ε, και θα πρέπει δηλαδή εδώ να βρεθεί μια ισορροπία που θα λαμβάνει υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία. Και έτσι πιστεύω πως θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή τη δικασία απλοποίησης. Νομίζω πως απάντησα σε όλες σας τις ερωτήσεις κύριε Νίκολσον ή όχι. James. Επερώτηση. Όχι, δεν απαντήσατε, αλλά ίσως και να σας υπέβαλα πολλές ερωτήσεις σε μια φορά. Εγώ αυτό που προσπαθώ να σας πω, κύριε υποψήφιε επίτροπε, είναι ότι επικρατεί απόγνωση στους ε, αγρότες σε όλα τα μήκη πλάτη της Ένωσης ένα σωρό παράπονα όσον αφορά την εισαγωγή προϊόντων που δεν παράγονται με τις ίδιε προδιαγραφέ και κανόνε όπω αυτοί που ισχύουν εδώ. Οι ε, γεωργοί τα έχουν βαρεθεί όλα αυτά. Δεν αντέχουν άλλο. Έχουν βαρεθεί και τη την γραφειοκρατία. Εντάξει, ορισμένε είναι ευθύνε των εθνικών κυβερνήσεων. Τι θα κάνετε για να του προκαλέσετε να, να, να, να αφαιρέσουν την γραφειοκρατία, να την καταργήσουν. Και ίσω να απαντήσετε και την άλλη ερώτησή μου που ήταν πώ ανακατανέμεται τους, ε, τα κονδύλια στους ενεργούς γεωργούς και τι είναι ακριβώς, τι ορίζεται ως ενεργός γεωργός, γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο μέλλον καθώς θα προχωρήσουμε, γιατί θα δημιουργήσουμε μια γεωργική, μια, γεωργική, μια αγροτική κοινωνία που να είναι βιώσιμη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Επίτροπε, απαντήστε. Ένας ενεργός ε, γεωργός είναι αυτός ο οποίος εγγυάται παραγωγή στοιχειώδη που έχει ε, έσοδα από την δραστηριότητά του και που έχει και τη δική του παραγωγή τροφίμων. Πράγμα που συνδέεται άμεσα με την επαγγελματική του παραγωγική δραστηριότητα. Από αυτή την άποψη, οι ενισχύσεις θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν αυτή τη κατάσταση. Έπειτα για τις προδιαγραφές και τους κανόνες που εφαρμόζουμε εδώ στην Ευρώπη. Εμείς δεν μπορούμε να επιβάλλουμε συγκεκριμένη νομοθεσία εκτός Ευρώπης. Δεν μπορούμε αυτά να τα επιβάλλουμε εκτός, ο, κυρίως όσον αφορά τις προσδοκίε των καταναλωτών σε σχέση με τη δική μας ε, γεωργία. Μπορούμε όμως ε, να ελέγξουμε τι εισαγωγές. Και τώρα, όσον αφορά την, τα ίδια τα κράτη-μέλη, με τον τρόπο τον οποίο θα συντάξουμε την ε, νομοθεσία μας, αυτή θα πρέπει να συνταχθεί χωρίς, όπως σα είπα, να αποδυναμώσει τις δυνατότητες ελέγχου και σωστή κατανομής των ε, ταμείων. Λέει η Αρίκα έχει τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Πίτροπε, εδώ βρίσκομαι. Η εμπειρία δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια η απορρίθμιση που έχει ξεκινήσει μας οδήγησε σε αποτυχία. Αποτυχία από όλες τις απόψεις. Δεν πιστεύετε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει μια πρωτοβουλία διεθνούς εμβέλειας ώστε να δηλώσει την ε, πράξη της γεωργικής παραγωγής ως μια αποστολή κοινοφελή με βάση το του μόλις. Δηλαδή μια αποστολή για την διατροφή, για την ανάπτυξη των εδαφών, ε, για το περιβάλλον δεν νομίζετε πως ο καλύτερος τρόπος να γίνει κάτι τέτοιο είναι να επανέλθουμε πραγματικά στις ε, ελάχιστες ενδοευρωπαϊκές τιμές οι οποίες ε, να είναι εγγυημένες, να μπορούσαμε να τις εγγυηθούμε για ένα συγκεκριμένο όγκο παραγωγής και θα μπορούσαμε από κοινού να αποφασίσουμε για το επίπεδο, ένα μέσο όγκο ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έπειτα για το θέμα των ενισχύσεων δεν θα πρέπει αυτές να ρυθμίζονται διαφορετικά δεδομένων όλων αυτών των αποστολών των Γεωργών. Επίτροπε. Κοιτάξτε κύριε Λαρίκα. Καταλαβαίνω απόλυτα τις, ε, ε, την ερώτησή σας σε σχέση με τη δυνατότητα του, Ευρωπαϊκού, του Ευρωπαίου Γεωργού να μπορέσει να θέσει σε εμπορία τα προϊόντα του. Αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και είναι αμφίδρομη. Δηλαδή προσφέρουμε πράγματα αλλά λαμβάνουμε κιόλα. Δηλαδή η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και αυτή η ανταγωνιστικότητα μας επιτρέπει αυτή τη στιγμή να είμαστε ένας από τους κεντρικούς, τους βασικούς εξαγωγούς ε, τροφίμων ακόμα και αν εισάγουμε επίσης. Δεν βλέπω λοιπόν πώ θα μπορούσαμε εκ νέου να χτίσουμε ένα φρούριο προστατεύοντα την εσωτερική μα αγορά. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η προστασία, οι εγγυημένε τιμέ δεν έχουν νόημα. Και γι' αυτό και η διαδικασία αποσύνδεση των ενισχύσεων γίνεται παράλληλα με το άνοιγμα των αγορών αλλά συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί ρύθμισης της αγοράς που θα διασφαλίζουν τουλάχιστον δύο πράγματα. Καταρχήν, σταθερότητα των εσόδων των γεωργών και δεύτερον, μια κάποια σταθερότητα των τιμών και πάλι θα πρέπει να αφήσουμε να παίξει και η προσφορά και η ζήτηση γιατί διαφορετικά φτάνουμε σε δημόσια στόκ τα οποία μας κοστίζουν πολύ ακριβά. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθούν οι λύσεις η λύση δεν είναι να πάμε πίσω, αλλά να προσπαθήσουμε να βρούμε νέους μηχανισμούς και αυτό να πιστεύω πως είμαστε σε θέση να το κάνουμε. Στη Γεωργία είναι ένα σημαντικό στοιχείο των διεθνών διαπραγματεύσεων αυτό, αλλά εδώ που συμφωνώ είναι ότι θα πρέπει ακόμα και μέσω αυτών των διαπραγματεύσεων να διασφαλίζουμε τις ικανότητες κάθε περιοφέρειας του κόσμου να μπορεί να αξιοποιήσει καταρχήν το δυναμικό της και τις ε, διεθνείς συναλλαγές, οι διεθνείς συναλλαγές να γίνονται με σεβασμό αυτής της αρχής. Ρίκ. Το κατανοώ αυτό που εξηγείτε, αλλά μέσα στη διεθνή πρωτοβουλία που θα μπορούσαμε να προτείνουμε και που φυσικά δεν θα γίνει εν μία νυχτή ούτε αναγκαστικά κατά τη διάρκεια της δικής, της δικής μας θητείας, μήπως θα μπορούσαμε να βρούμε παρόμοιους μηχανισμούς ε, παροτρύνοντας ε, τις άλλες υπήρους ή τις άλλες ομάδες χωρών ε, να κάνουν το ίδιο όπως και εμείς, πράγμα που θα είχε το πλονέκτημα να εγγυηθεί την τροφική κυριαρχία όλων. Ναι, βεβαίως. Πιστεύω ότι σεβόμενοι αυτή την αρχή, σεβόμενοι τις αρχές του διεθνούς εμπορίου, και ξεκινώντας με βάση αυτές τις αρχές της πολυ πολικής οικονομίας των διαφόρων περιφερειών, ότι δηλαδή μπορούμε να έχουμε περιφέρειες με ε, ομοιογενείς ε, ανταγωνιστικές δυνατότητες. Εγώ είμαι έτοιμος να στηρίξω αυτού του είδους τις ιδέες, αλλά και πάλι να πω χωρίς απόλυτη απομόνωση των αγορών, γιατί πιστεύω πως αυτό δεν είναι εφικτό και δίνοντας τη δυνατότητα στις διάφορες περιφέρειες του κόσμου να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους και να υπάρχει εμπορική, να γίνονται ισότιμες ε, εμπορικές συναλλαγές. Από αυτή την άποψη μπορείτε να βασίζεστε σε μένα. Είναι ο, η σειρά του Τζαν Κάρλο Κοτά. <clears throat> Ευχαριστώ τον κύριο Τσόλος ε, για την ε, παρουσία του. Τα ζητήματα που ετέθησαν είναι πολύ σημαντικά. Αυτό όμως που θέλω να το ρωτήσω εγώ είναι η ανάπτυξη της υπαίθρου και πιο συγκεκριμένα η ανάπτυξη των πιο μειονεκτικών περιοχών, ορεινών περιοχών ας πούμε. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει προς τη θέμηνη αξία για την οικονομική και δημογραφική ανάπτυξη για τις μειονεκτικές περιοχές και εγώ που έρχομαι από το Πιεμόντε θέλω να ρωτήσω πώς θα αναζωογονήσετε τις εγκαταλελειμμένες γεωργικές περιοχές οι οποίες δημιουργούν υποβάθμιση όχι μόνο περιβαλλοντική αλλά και κοινωνική και την έχουν όλοι μπροστά στα μάτια τους, την βλέπουν όλοι. Ο δεύτερος πυλώνας της ε, ΚΑΠ επιτρέπει με το ειδικό μέσο στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες να εφαρμόσουν ειδικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Εγώ φυσικά στη διάρκεια της εντολής μου και όσο θα προχωράει η εντολή μου ελπίζω η ΚΑΠ μετά το 2013 θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να έχουν περισσότερα μέσα στη διάθεσή τους για αυτές τις περιφέρειες και πιο συγκεκριμένα τις μειονεκτικές περιφέρειες των οποίων θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε το τοπικό δυναμικό. Πιστεύω λοιπόν ότι η συνεργασία θα πρέπει να αναπτυχθεί σε τοπικό επίπεδο με την ανάπτυξη δικτύων ε, στην ε, γεωργία και στους άλλους τομείς της ανάπτυξης της υπαίθρου. Ο δεύτερος πυλώνας μας δίνει αυτή τη δυνατότητα και στον πρώτο πυλώνα τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα ανάλογα με την οικονομική ευρωστία της ΚΑΠ τα κράτη-μέλη μπορούν να απαντούν ενισχύοντας τους πιο αδύναμους τομείς στη Γεωργία που υποφέρουν. Ο Τζαν και πάλι. Σύντομη απάντηση. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Γεωργία είναι η απομίμηση των γεωργικών προϊόντων. Το κοινοτικό καθεστώς προβλέπει τα προστατευμένα προϊόντα ε, γεωγραφικής προέλευσης. Εσείς τι μέτρα θέλετε να λάβετε ούτως ώστε να πατάξετε την απομίμηση αυτών των προϊόντων. Εγώ θέλω να προστατεύσω τα προϊόντα τα οποία είναι ντόκ ή έχουν ειδική γεωγραφική προέλευση. Θέλω λοιπόν να αναδαφνίσω τις οδηγίες που αφορούν την ποιότητα δηλαδή τα ντοκ, τα ΙΖΕΠ και τα λοιπά, για να μπορέσουμε, ονομασίες δηλαδή προέλευσης ή γεωγραφικής προέλευσης, για να μπορέσουμε να βρούμε τα στοιχεία της ποιότητας που θα προβάλλουν αυτά τα προϊόντα. Για παράδειγμα, εγώ σκέφτομαι, έχω κατά νου δηλαδή τώρα το ελαιόλαδο, να βρούμε νέες τεχνολογίες, νέους μηχανισμούς που θα μας επιτρέπουν να ελέγχουμε καλύτερα την αγορά και όλες αυτές τις απάτες οι οποίες διακυδεύουν το εμπόριο αυτών των ευρωπαϊκών προϊόντων ποιότητας. Ό,τι περνάει λοιπόν από το χέρι της Επιτροπής ρυθμιστικά θα το κάνουμε. Ελπίζουμε και οι παραγωγοί να κάνουν και αυτοί τις προτάσεις τους όταν πρόκειται για τοπικό προϊόντα. Για την Άλντε, η κυρία Ρέμερς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και η Άλντε σας καλωσορίζει εδώ σήμερα κύριε Σιόλος. Σας ρωτώ ως φιλελεύθερη το εξή. Η ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική και τα προϊόντα της έχουν πολύ υψηλή ποιότητα αλλά και υψηλό κόστος. Για στον αγώνα κατά των χωρών που παράγουν φτηνά σας ερωτώ πώς μπορείτε με τρόπο συμβατό προς τον ΠΟΕ να προάγεται τα προϊόντα μας. Ποιους μηχανισμούς έχετε συγκεκριμένα υπόψη και ως ε, αγρότης σας ε, ρωτώ τι διασφαλίζει καλύτερα τους αγρότες. Να αφιερώσουμε χρόνο για να διασφαλίσουμε την παραγωγή μας ή να πιστοποιήσουμε την παραγωγή αυτή. Απάντηση ο Επίτροπος. Ναι, το είπα και στην εισαγωγή μου. Τα ειδικά χαρακτηριστικά της γεωργικής παραγωγής σχετίζονται και με, την, με τα υψηλά ποιοτικά πρότυπα των προϊόντων μας. Αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί και στις διεθνείς αγορές, δηλαδή και στις διεθνείς επραγματεύσεις, αλλά πολύ ιδιαίτερα και στην προώθηση των προϊόντων και σκοπεύω να προτείνω σχετικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν μπορώ να πείσω τους Ευρωπαίους εταίρους μας ότι από κοινού μπορούμε να δράσουμε καλύτερα και να ε, ασκήσουμε καλύτερη εμπορία σε παγκόσμιο επίπεδο, θα είμαι ευτυχής. Υπάρχουν διαφορετικές αγορές και διαφορετικές ε, δυνατότητες ε, πώλησης στις αναπτυσσόμενες χώρες ε, υπάρχει όλο και μεγαλύτερη τάση για ασφαλή προϊόντα σιγά σιγά. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το δυναμικό να το αξιοποιήσουμε ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα προϊόντα μας και την ε, ασφάλεια των προϊόντων μας. Αυτό εξαρτάται από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται. Αυτά τα πρότυπα λοιπόν είναι πολύ σημαντικά. Θα πρέπει και να τα κάνουμε γνωστά, αλλά και να τα προωθήσουμε για να γνωρίζει ο καθένας τι σημαίνει ακριβώς αυτή η ποιότητα την οποία και ενισχύουμε, αλλά και ο τομέας, ο κλάδος των τροφίμων έχει σημαντικό ρόλο να διδραματίσει για να αντισφαλίσει αυτή την ποιότητα των τροφίμων. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντική και η συνεργασία μεταξύ των παραγωγών, των μεταποιητών, των, των εμπόρων. Δεν είναι σημαντική δηλαδή μόνο οι μηχανισμοί, και η ενίσχυση των προϊόντων μας, η πρόθεση των προϊόντων μας, γιατί θέλουμε ιδιαίτερα να προωθήσουμε ιδιαίτερα σωστά προϊόντα, αλλά είναι υπεύθυνοι και αυτοί οι οποίοι τελικά είναι οι μεταποιητές των προϊόντων. Η επόμενη ερώτηση. Αν δεν θέλετε λοιπόν άλλη ερώτηση. Να περάσουμε λοιπόν ε, στον συνάδελφο Μόρβεϊ, στην κυρία Μόρβεϊ. Köszönöm szépen, itt vagyok, elnök úr, és magyar σας ευχαριστώ εδώ είμαι. Θα ήθελα να ρωτήσω, να θέσω το ερώτημά μου στα ουγγρικά. Υποψήφιε επίτροπε, είσαστε, είσαστε υποψήφιος από τη Ρωμανία και συνειδητοποιείτε ότι λοιπόν οι, προ... πρώην κομμουνιστικές χώρες, στις πρώην κομμουνιστικές χώρες, η Γεωργία έχει περάσει ακόμα πιο βαθιά κρίση από όλη την υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη. Και οι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι μικρές επιχειρήσεις, ήταν αυτές που τελικά αντιμετώπισαν τα πιο μεγάλα προβλήματα. Και πλέον απειλείται η επιβίωσή τους. Θα ήθελα να διαθέσετε τα δύο λεπτά που έχετε στη διάθεσή σας για να μας πείτε πώς σκοπεύετε να βοηθήσετε τις μικρές ε, και οικογενειακές επιχειρήσεις και γιατί θα πρέπει να σας ψηφίσω αν θέλω να υποστηρίξω αυτές τις επιχειρήσεις. Παρακαλώ να είστε συγκεκριμένος. Απάντηση. Οι μικρές ε, επιχειρήσεις αποτελούν πάρα πολύ σημαντικό τμήμα του συνόλου των επιχειρήσεων για τα νέα κράτη-μέλη και όχι μόνο για τα νέα κράτη-μέλη αλλά και για τα παλιά κράτη-μέλη κυρίως ε, και στην ε, Νότια Ευρώπη βλέπουμε να επαναλαμβάνεται αυτό το πατρόν. Χρειαζόμαστε λοιπόν μία πολιτική εξυγχρονισμού και νομίζω ότι ο δεύτερος πυλώνας της ΚΑΠ θα πρέπει να διαμορφωθεί με τρόπο τέτοιο προκειμένου για να προσαρμοστεί στις μικρές, στα χαρακτηριστικά αυτά των μικρών επιχειρήσεων και θα πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Να εξυγχρονίσουμε τις εκμεταλλεύσεις και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα του δεύτερου πυλώνα. Όχι απαραίτητα για να καταστούν πιο μεγάλες αν θέλετε, αλλά για να εξυγχρονιστούν να προσφέρουν πιο ποιοτικά προϊόντα στις σύγχρονες αγορές. Αυτό που ως τώρα δεν έχει ακόμα αξιοποιηθεί ιδιαίτερα είναι οι τοπικές αγορές, οι οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν περισσότερο. Αυτές οι μικρές επιχειρήσεις δεν χρειάζονται να παράγουν για εξαγωγές. Το βλέπω και στη χώρα μου και σε άλλες χώρες. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για συγκεκριμένα τοπικά, παραδοσιακά προϊόντα. Και θεωρώ ότι σε αυτά τα προϊόντα, σε αυτές τις αγορές θα πρέπει να επικεντρωθούν οι μικρές επιχειρήσεις, οι μικρές εκμεταλλεύσεις. Και θα ήθελα να χρησιμοποιήσω ακριβώς τα μέσα του δεύτερου πυλώνα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και του πρώτου πυλώνα. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και σας λέω ότι πέρα από, τα, από τις θα πρέπει να συνεχιστεί το πρόγραμμα μεταρρύθμισης και η προσαρμογή στις τοπικές αγορές. Ναι, χάρηκα που άκουσα ότι είπατε ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην τοπική παραγωγή, στις τοπικές αγορές. Πώς θα γίνει αυτό, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τις ίδιες μας τις αγορές από την ε, υπερβολική επιδότηση ξένων προϊόντων, τα οποία συχνά είναι και χαμηλή ποιότητα. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα μέτρα τα οποία σκοπεύετε για τα μέτρα που σκοπεύετε να λάβετε τους επόμενους 12 μήνες, για παράδειγμα, για να βοηθήσετε τους μικρούς αγρότες στη Ρουμανία, στην Ουγγαρία. Δηλαδή, αν παρακολουθήσουμε την ακρόαση αυτή σε ένα χρόνο, τι θα μπορέσουμε να πούμε, ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Απάντηση. Ναι. Μπορούμε θεωρώ να το πετύχουμε αυτό με τις προτάσεις για την ΚΑΠ μετά το 2013. Κατά τη διάρκεια του έτους αυτού λοιπόν θα γίνει μια συζήτηση και μέχρι τα τέλη του 2010 σκοπεύω να δημοσιεύσω μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για προτάσεις σχετικά με την μελλοντική ΚΑΠ και ελπίζω εκεί να βρείτε και νέες προτάσεις για το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο και την διαδικασία της συζήτησης αυτής, δεν θα είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα λάβει τις αποφάσεις. Θα συμμετάσχουν και άλλοι φορείς και Επίσης, στην Επιτροπή σας υπάρχουν πολλές ιδέες για την ε, μεταρρύθμιση της κατάστασης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως σε ό,τι αφορά τις προμήθειες σε τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω δυνατότητες, γιατί αποτελούν σημαντικό α, τμήμα της ενιαίας αγοράς. Και σίγουρα θα μπορέσουν να συμπεριληφθούν στις προτάσεις αυτές για την διαμόρφωση της ΚΑΠ μετά το 2013. Andiamo Τελειώσαμε τον πρώτο γύρο, πάμε στο δεύτερο. Εγώ θέλω να σας υπογραμμίσω ότι δεν εξοικονομήσαμε ούτε ένα λεπτό. Με εξαίρεση την Άλντε, γιατί έχουμε ένα σημαντικό αριθμό βουλευτών που θέλουν να τοποθετηθούν. Στους, σε αυτόν τον επόμενο κύκλο ε, τοποθετήσεων σας παρακαλώ εξοικονομήστε χρόνο. Ο κύριος Παπαστάνκος. How do you assess Ευχαριστώ, Πρόεδρε Δεκάστρο. Κύριε Τσιόλος, πώς ε, αποτιμάτε τις πιθανές, ε, τον πιθανό αντίκτυπο στην ε, Ευρωπαϊκή Γεωργία της των διατυπώσεων που συμφωνήθηκαν στον ΠΟΕ τον Ιούλιο του 2008 και των μετέπειτα προσαρμόσεων που θεωρείται ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση θα πρέπει να τηρήσει την ήδη υπό εξέλιξη μεταρρύθμιση την προϋπόθεση ότι θα πετύχουμε τις αντίστοιχες ε, υποχωρήσεις και δεσμεύσεις και από τους εμπορικούς μας εταίρους. Σας ευχαριστώ. Με αυτή την άποψη πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει πολύ συνεπείς προτάσεις σε σχέση με τη Γεωργία και τώρα θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι προτάσεις που θα μας υποβάλουν οι εταίροι μας. Εμείς θα πρέπει να είμαστε πολύ σταθεροί στις απόψεις μας. Ήδη σε ευρωπαϊκή κλίμακα κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια, ιδιαίτερα όσον αφορά την, ε, το άνοιγμα της αγοράς μας. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πέρα από τα όσα ήδη παρουσιάσαμε. Έχουμε κάνει πρωτοβουλίες, θέλουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία ώστε όλα τα μέρη να μπορέσουν να βγουν κερδισμένα. Μια πολυμερή συμφωνία. Ωστόσο τώρα θα πρέπει εμεί να περιμένουμε να δούμε ποιε θα είναι οι αντιπροτάσεις των εταίρων μας. Γιατί οι δικές μας προσπάθειες ήδη ήταν σημαντικέ, Γιώργο. Οι the recent uh, agreements uh, γεωργική αναταχή με τις μεσογειακές χώρες και όχι μόνο απέδειξαν ότι το άνοιγμα της αγοράς χωρίς ε, ρυθμιστική ισορροπία δημιουργεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα στους δικούς μας παραγωγούς. Πώς προτίθεστε να ενσωματώσετε καλύτερα τις ε, μη ε, τα, τους μη εμπορικούς προβληματισμούς στις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ περί Γεωργίας σε σχέση με την πολυλειτουργική ε, τον πολιτικό χαρακτήρα της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρείται πως θα είναι επιτυχές αποτέλεσμα στις γεωγραφικές ενδείξεις θα είναι ένα ουσιώδες τμήμα μιας, ισορροπη... ενός, μιας ισορροπημένης συμφωνίας στο ΠΟΕ περί γεωργίας. Επίτροπε. να σας πω. Αν αναφέρεστε στο πακέτο για τις γεωργικές ενδείξεις, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να φτάσουμε σε συμφωνία, γιατί αυτό το στοιχείο αποτελεί τη βάση της ε, πολιτικής του, γεωργο, του γεωργοδιατροφικού τομέα της Ευρώπης. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να εστηρίζουμε το μοντέλο αυτό και να ελπίζουμε πως οι εταίροι μας θα το αναγνωρίσουν και ότι θα αποδεχτούν ότι τα δικά μας προϊόντα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, ε, των διαπραγματεύσεων. Οι γεωγραφικές ενδείξεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των διαπραγματεύσεων για μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να πω, Πρόεδρε, ότι με τις απάντησεις του κυρίου Τσιόλου σήμερα μπορούμε να σιγουρευτούμε ότι αυτό το μη έγγραφο έχει πάει στα σκουπίδια και συμβουλεύω να μην πάει να το ψάξει κανείς, καλά θα κάνει το αφήσει εκεί που είναι. Σε όλες τις απαντήσεις που δώσατε ήσασταν σαφέστατος ε, για τον πρώτο και το δεύτερο πυλώνα. Πρώτος πυλώνας με τις ε, αποζευγαρωμένες ε, ε, ενισχύσεις συγγνώμη, και μετά τον δεύτερο πυλώνα με την ανάπτυξη της υπαίθρου της μικρές εκμεταλλεύσεις. Μήπως όμως εσείς έτσι μας εγκλωβίζετε σε δύο τύπου γεωργίες, αυτές δηλαδή που ενισχύονται από τον πρώτο πυλώνα, από, ενισχύονται από το κράτος και τη δεύτερη κατηγορία η οποία θα κάνει ανάπτυξη της υπαίθρου και άλλα πράγματα. Εγώ προτείνω να έχουμε μία συνολική γεωργία η οποία να είναι και κατανοητή από τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτοί οι δύο πυλώνες είναι γρίφος για τους πολίτες. Ναι, εγώ γνωρίζω και τις σκέψεις σας και τις ανησυχίες σας σχετικά. Εγώ δεν είμαι κλεισμένος ως προς τη μορφή πρώτος πυλώνας, δύο πυλώνες. Αυτό το οποίο έχω σήμερα εγώ κατά νου είναι η ουσία. Και όχι, είναι το περιεχόμενο και όχι η μορφή. Δηλαδή οι δύο πυλώνες μπορούν να αναφέρονται σε σε όλες τις γεωργίες που ανέφερα, γιατί έχουμε πολλές γεωργίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν εμείς έναν πυλώνα, εμείς δεσμευτούμε σε μία αιτήσια ε, βάση πληρωμών, ε, διότι έχουμε εξάλλου διατάξεις ε, περιβαλλοντικού χαρακτήρα κλπ. Ήδη και ο δεύτερος πυλώνας θα επέτρεπε να εξυγχρονιστούν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις ε, διότι οι αλλαγές του κλίματος θα μας επιβάλλουν αυτόν τον εξυγχρονισμό. Μία καλύτερη σύνδεση μεταξύ γεωργίας και υπαίθριου χώρου. Βεβαίως και μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε πολιετής ε, ε, προγραμματισμούς και μπορούμε να προβληματιστούμε γύρω από αυτά τα προγράμματα. Εγώ λοιπόν δεν είμαι ε, αμετάκλητος ως προς τη μορφή σε αυτή τη φάση αλλά ε, για το περιεχόμενο επιμένω Εξαλλού και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την ήδη υπάρχουσα νομοθεσία και να τη χρησιμοποιήσουμε για να εξυγχρονιστούμε και για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ Επίτροπε ο Στεφάν. Ναι εντάξει άκουσα την απάντηση. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι θα μας επιτρέψει να συζητήσουμε για την γεωργική πολιτική, τους γεωργούς, την κοινωνία και την Ευρώπη συνολικά είναι το να καταστήσουμε ε, κατανοητή την ΚΑΠ από τον πολίτη. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα εγώ, δηλαδή, πρώτος πυλώνας, όχι συγχρηματοδότηση, ο δεύτερος πυλώνας, συγχρηματοδότηση. Αλλά όμως ορισμένα κράτη ε, σμπρώχνουν στη σύγχρηματοδότηση και για τους δύο πυλώνες η θέση μου είναι η εξής. Όταν έχουμε μία ΚΑΠ, ε, τότε αφού είναι κοινή αγροτική πολιτική θα πρέπει να έχουμε και έναν κοινό προπολογισμό. Ε, για την ανάπτυξη της υπαίθρου η συγχρηματοδότηση έχει, παίζει ένα διαφορετικό ρόλο από αυτόν του πρώτου πυλώνα. Πάντως σε αυτή τη φάση αυτή είναι η θέση μου. Χρειαζόμαστε κοινοτικό προϋπολογισμό για τις ε, κοινοτικές ε, πολιτικές. Και φυσικά δεν θα πρέπει εμείς ε, να απαγορεύσουμε την ενίσχυση σε κρατικό επίπεδο ο Λάιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά, να σα ε, ζητήσω συγγνώμη που καθυστέρησα, καθυστέρησε πτήση από το Εδιμβούργο. Να σας ρωτήσω ποιες είναι τα, ποια είναι τα τρία μέτρα τα βασικά τα οποία είναι πιο σημαντικά και θα λάβετε τα επόμενα χρόνια για να προωθήσετε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Μισάριο. Yes, very briefly, I think that... Εν συντομία, νομίζω ότι καταρχάς η προσαρμογή της ε, κοινή αγροτικής πολιτικής θα κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή για να αυξήσει ακριβώς την ανταγωνιστικότητα και νομίζω ότι τα μέτρα τα επενδυτικά και η προσαρμογή των ε, γεωργών στις καινούργιε αυτές συνθήκες θα είναι σημαντικές γιατί οι προσαρμογές αυτές δεν ε, θα μειώσουν απαραίτητα την ανταγωνιστικότητα, άρα επενδύσεις για τον εξυγχρονισμό. Και θεωρώ ότι στον πρώτο πυλώνα ο τρόπος που θα ισορροπήσουμε τις άμασες πληρωμές θα μπορέσει και αυτός να συνεισφέρει προς αυτή την κατεύθυνση και στις διεθνείς διαπραγματεύσεις νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε στα αποτελέσματα που θα πετύχουμε στους αγρότες μας τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν καλύτερα τις διεθνείς αγορές. Με τα αποτελέσματα που θα πετύχουμε δηλαδή, να δώσουμε νέες ευκαιρίες στους αγρότες μας. Νομίζω ότι αυτά θα είναι τρία βασικά στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να τα προασπίσουμε, αλλά και να τα εφαρμόσουμε για να προωθήσουμε την ανταγωνιστικότητα. Τζόρτς, ναι, άκουσα τι είπατε θα σκεφτείτε κάποια από τα νέα βιοτεχνολογικά εργαλεία τα οποία έχουν στη διάθεσή του αγρότες ε, στον υπόλοιπο κόσμο. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά και οι Ευρωπαίοι αγρότες. Μπορεί να πείτε ότι δεν εντάσσεται αυτό στο χαρτοφυλάκιό σας, αλλά αποτελεί σημαντικό θέμα για, την, ε, για τον κλάδο. Αν θα μπορούσατε λοιπόν να μας πείτε ποια είναι η στάση σας και τι δράση θα αναλάβετε στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να διασφαλίσετε ότι οι αγρότες μας θα έχουν ακριβώς την διαπρόσβαση στα ίδια εργαλεία όπως και οι αγρότες στον υπόλοιπο κόσμο. Απάντηση. Μιλήσατε για την ανταγωνιστικότητα. Νομίζω ότι για να είναι κανείς ανταγωνιστικός στη γεωργία θα πρέπει να έχει πελάτες, να έχει καταναλωτές. Άρα, σε ό,τι αφορά την βιοτεχνολογία, νομίζω ότι είναι απαραίτητο στην εσωτερική αγορά να πείσουμε τους καταναλωτές ή τέλο πάντων να δώσουμε την ευκαιρία στον καταναλωτή να κάνει την επιλογή του. Θέλει ή δεν θέλει προϊόντα με γενετικά τροποποιημένου οργανισμούς. Αλλά φυσικά εξαρτώμαστε και από τις αγωγές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ζωοτροφές. Και άρα προς την κατεύθυνση αυτή θεωρώ ότι στο νέο σώμα των επιτρόπων θα πρέπει να βρεθούν λύσεις για να δοθεί στους εκτροφείς ζώων δυνατότητα να αναπτύξουν την δραστηριότητά τους, να μην ε, τους πλήξει αυτό το πρόβλημα λόγω της ρύθμισης, άρα και τις βιοτεχνολογίες, νομίζω ότι είναι σημαντικό. Είναι ένα σημαντικό επιστημονικό επίτευγμα προς την κατεύθυνση αυτή και μετά θα πρέπει να δούμε πώς θα πείσουμε τους καταναλωτέ να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα αυτά. Γιατί για την κοινή μας ενιαία αγορά θεωρώ ότι είναι βασικό αυτό στο ευρύτερο πλαίσιο της ποιοτική πολιτικής, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη και τον παράγοντα του καταναλωτή. Μάλιστα. Και τώρα ο Ζωζέ Μποβέ. Κύριε Επίτροπε, καλημέρα. Θα ήθελα να συνεχίσω γύρω από αυτό το θέμα. Ακούσατε μία γνώμη. Αλλά Δείτε πού βρισκόμαστε με το πρόγραμμα Coextra. Δείτε τι γίνεται σήμερα με τη συνύπαρξη μεταξύ παραγωγής και του δικτύου γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, μη γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Πώς μπορούμε εμείς να εγγυθούμε την ελευθερία επιλογής και για τους αγρότες αλλά και για εκείνα τα γεωργικά δίκτυα τα οποία θέλουν να εγγυηθούν μία διατροφή χωρίς γενετικά τροποποιημένου οργανισμούς. Και φυσικά εδώ όπως το υπογραμμίσατε έχουμε και το πρόβλημα που συνδέεται με τις εισαγωγές, τις εισαγωγές της σόγιας. Σήμερα ο περιορισμός σε περιεκτικότητα ε, φυτικής ε, πρωτεΐνης ε, περιορίζει την εισαγωγή αυτών των προϊόντων. Αλλά πώς ενισχύονται εκείνα τα δίκτυα τα οποία θα ήθελα να παράγουν χωρίς γενετικά τροποποιημένες ουσίες. Εγώ συμφωνώ. Συμφωνώ ότι ο καταναλωτής πρέπει να μπορεί να διαλέγει για προϊόντα με ή χωρίς γενετικά τροπημένους οργανισμούς. Δεν θέλω να αποφύγω την απάντηση, αλλά αυτό ξέρετε ότι είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία είναι αρμόδια για να αποφασίσουν για το κατά πόσο θα συνεπάρχουν αυτές οι δύο μέθοδοι παραγωγής. Πρόκειται λοιπόν, είπα, για εθνική αρμοδιότητα. Τώρα, για τη φυτική πρωτεΐνη, τη σόγια πιο συγκεκριμένα σήμερα, με τους διεθνείς εμπορικούς κανόνες, εμείς δεν δεσμευόμαστε στο να περιορίζουμε την η καλλιέργεια διότι εμείς έχουμε αποσυνδέσει τις ε, ε, ενισχύσεις δεν μπορούμε στην προκειμένη περίπτωση να τις ε, ξανασυνδέσουμε και ορισμένα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα, την κλιματική δυνατότητα να καλλιεργούν σόγια Θα πρέπει λοιπόν εμείς να δούμε πώς μπορούμε να ισορροπήσουμε την κατάσταση διότι σε αυτές τις καλλιέργειες δεν θα φτάσουμε ποτέ σε αυτάρκεια και εντάξει μπορούμε εμείς να φυτέψουμε και να καλλιεργήσουμε καλαμπόκι ή σόγια αλλά τίποτα δεν μας απαγορεύει να εισάγουμε το κρέα ζώων που τράφηκαν με αυτά τις ουσίες. Τώρα εγώ πιστεύω, λέει ο κύριος Μποβέ, ότι θα μπορέσουμε στο μέλλον να συνεργαστούμε με την Κομισιόν για αυτά τα θέματα. Εσείς μιλήσατε για την ποιότητα, είναι πολύ σημαντικό για μένα. Σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει μία κάπως σκανδαλώδης κατάσταση και ο νέος επίτροπος ελπίζω ότι θα πρέπει να ξαναρχίσει τη συζήτηση με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Πώς μπορούμε εμείς να δεχτούμε όταν έχουμε ήδη ρυθμίσει τον πόλεμο για τα βοηδή με ορμόνες για τρία χρόνια ακόμα η Ευρώπη υπερφορολογεί 100% ενώ έχει λήξει το πρόβλημα. Πρέπει να σταματήσει λοιπόν η Κομισιόν αυτό το διεθνές σκάνδαλο. Ναι, καταλαβαίνω τις ανησυχίες σας. Οι διεθνεί διαπραγματεύσει είναι αρμοδιότητα του συναδέλφου μου Κάρελ Ντεγκούχτ και εγώ είμαι έτοιμος να συνεργαστώ μαζί του για να δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα διότι εκκρεμεί εδώ και πολύ καιρό. Ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε μία λύση γι' αυτό. Ο, κύ, ο κύριος Χάσγουρτ. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίτροπε, νομίζω ότι θα πρέπει να διερευνήσουμε τις απόψεις για ανακατανομή λίγο περισσότερο. Εγώ με την άποψή σας ότι πρέπει να απομακρυνθούμε από την ιστορική βάση, ότι πρέπει να βρούμε νέες λύσεις. Θα ήθελα να προτείνω ότι οι αρχές για τα νέα κριτήρια στήριξης θα πρέπει να είναι απλούστερα, δεύτερον θα πρέπει να είναι πιο ισότιμα και δεύτερον πιο ε, διαφανή. Υπάρχει άποψη σε διάφορα έθνη και ιδιαίτερα τονίζω μεταξύ των νέων ε, κρατών μελών ότι οι ισοπεδωμένα ποσοστά με βάση την εκτάσεις φαίνεται να είναι μια λογική εξέλιξη. Πιστεύετε πως έχουν δίκιο? Σε σχέση με την κατανομή, νομίζω πως αναφέρεστε στην κατανομή στην τροφική αλυσίδα. Όχι, μίλησα για στήριξη της γεωργικής βιομηχανίας, δίκαιη και διαφανής. Προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω πως ήμουν αρκετά σαφής για την μελλοντική γεωργική πολιτική. Πιστεύω πως τα κριτήρια κατανομής των άμεσων πληρωμών θα πρέπει να αναλυθούν εκ νέου και να λάβουν καλύτερα υπόψη ορισμένα ειδικά στοιχεία που θα οδηγήσουν σε καλύτερη ισορροπία, ισορροπία επ' Ε, Επίσης, συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει ε, να υπάρχει ισότητα, δικαιοσύνη, είναι μια λέξη που χρησιμοποίησα, και η διαφάνεια. Τώρα η Επιτροπή ήδη έχει λάβει κάποια μέτρα για να είναι πιο διαφανή όσον αφορά την κατανομή αυτών των ενισχύσεων. Ε, οπότε τώρα νομίζω είναι θέμα της Κομισιόν σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο να αναλύσει τι θα χρησιμοποιήσει τελικά, να είναι απλούστερα τα κριτήρια, να είμαστε βέβαιοι πως τα ευρωπαϊκά χρήματα χρησιμοποιούνται σωστά. Ε, επίσης, ότι τηρείται η συμμόρφωση προς τα κριτήρια, ε, δικαιοσύνη και διαφάνεια. Ε, τα κράτη-μέλη να έχουν ήδη τη δυνατότητα να δώσουν μεγαλύτερη διαφάνεια, περισσότερη διαφάνεια στο επίπεδο των ενισχύσεων που λαμβάνουν κάποιοι γεωργοί. Έχω σκοπό λοιπόν να ακολουθήσω αυτή την κατεύθυνση. Επερώτηση. Ναι, Επίτροπε, συγκεκριμένα σας ρώτησα για τις απόψεις για τα, την βάση της επίπεδης ενίσχυσης επί τη βάση των εκταρίων. Αλλά πέρα από αυτό θα, θα απαιτηθούν και διορθωτικοί δημοσιονομικοί μηχανισμοί για το μέλλον. Ποια είναι η άποψή σας για αυτούς. Και βέβαια εδώ έχω κυρίως υπόψη μου την έκπτωση. το η επίπεδη ενίσχυση ανάμεσα με τα Ήδη υπάρχει ο μηχανισμός, ήδη έχει αποφασιστεί ότι θα περάσουμε σε μια ενίσχυση ανά εκμετάλλευση και θα, θα βασιστεί αυτή η ενίσχυση με ομοιόμορφο τρόπο και με βάση τις ενισχύσεις που είχαν ήδη λάβει οι, οι γεωργοί. Δηλαδή ενίσχυση με βάση εκτίμηση των προηγούμενων ενισχύσεων για τα παλιά κρατημέλη και επίπεδο ποσοστό ενίσχυσης με βάση τα εκτάρια για τα νέα κρατημέλη για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερη ισότητα στην κατανομή των ενισχύσεων. Ο κύριος Άγνιου. Όχι, τελειώσατε τώρα. Ο κύριος Άγνιου. Ευχαριστώ. Οι Βρετανοί παραγωγοί αυγών σε κλοβού αναγκάστηκαν πρόσφατα να αλλάξουν τα στήματά τη και η Ευρωπαϊκή Ένωση απογόρευσε την κυβέρνηση να δώσει βοήθεια. Από την άλλη πλευρά, η αντίστοιχη παραγωγή τη Ρουμανία επιτράπηκε να πάρουν βοήθεια και 25% από την Ένωση. Τμήμα των χρημάτων αυτών πληρώθηκαν από Βρετανού φορολογούμενου. Αν οι Ρουμάνοι αποφασίσουν να μην συμμετέχουν εκεί, συνεχίζουν να παράγουν σε κλοβού, σε συστοιχίε μετά από την απαγόρευση, ενώ οι Βρετανοί όχι. Τώρα, το να προεδρεύει ένας Ρουμάνος, Ρουμάνος επίτροπος εδώ μπορεί να θεωρηθεί ως υπερβολικό. Οι Βρετανοί φορολογούμενοι συμβάλλουν ε, στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Το 2002 δεπανήθηκαν πολύ άσχημα τα χρήματα του 2002. Εσείς θα εξυπηρετήσετε την ε, γαλλική σας, ε, τους γαλλικούς σας συνδέσμους και αν τελικά η ΚΑΠΑ στη Βρετανία αποδειχθεί καταστροφική θα τη σταματήσετε. Επίτροπε. Δεν κατάλαβα. σε ποια ενίσχυση αναφέρεστε. Το 2002 δεν ήμασταν μέλη της Ένωσης. Δεν ξέρω για ποια ενίσχυση μιλάτε λάβαμε κάποια ενίσχυση για τον εξυγχρονισμό του ε, αγροτροφικού τομέα, αλλά άλλο είδους ενισχύσεις δεν βήραμε γιατί η Ρουμανία δεν ήταν ακόμα κράτος μέλος της Ένωσης. Μπορείτε να διευκρινίσετε κάπως καλύτερα σε ποια κονδύλια αναφέρεστε, σε ποιους τομείς και σε ποια μέσα της ε, πολιτικής αναφέρεστε. Άγνιου. Κοιτάξτε, ήταν δύο χωρί τέσσερα. Μία αφορά το παρόν, που είναι η πιο σημαντική, και θέλω να επανέλθω γενικότερα, αν μου επιτρέπετε. Θέλετε να ολοκληρώσετε τα δύο λεπτά σας. Μα είχατε τη δυνατότητα να μιλήσετε για δύο λεπτά. Να σας τα πω γενικότερα για αυτά την απαγόρευση χρήση στοιχειών για την παραγωγή αυγών. Ιταλία και Ισπανία έχουν μείνει πίσω στην αλλαγή οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να τρώνε αυγά. Αλλά αν περάσει αυτή η απαγόρευση θα εισαχθούν από την Ινδία και από την Ουκρανία τα αντίστοιχα μέσα. Εκεί θα εισάγονται αυγά τα οποία παράγονται στην Ινδία και στην Ουκρανία και επίσης από κότε που έχουν τραφεί με διαφορετικό τρόπο από ό,τι αυτός που επιτρέπεται στην Ένωση. αναφέρεστε σε εκείνο τον κανονισμό που αφορά τις στοιχείες κλοβών. Εκεί προβλέπονται επενδύσεις για το τομέα. Αυτό έχει να κάνει με ε, την ευημερία των ζώων και ισχύει για όλους τους παραγωγούς, είτε είναι Βρετανοί είτε είναι Ρουμάνοι. Θα πρέπει να σεβαστούν αυτές τις διατάξεις. Εν πάση περιπτώσει, εγώ από όσο γνωρίζω, αυτοί οι κανόνε και η εφαρμογή του ήδη έχει ξεκινήσει. Υπάρχουν βέβαια μεταβατικές περίοδοι, οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται. Και Τόσο στη Ρουμανία όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει δυνατότητα στήριξη με συγκεκριμένε επενδύσει για τον εξυγχρονισμό του τομέα. Ελπίζω πω οι παραγωγοί θα μπορέσουν να σταθούν στο ύψο των περιστάσεων και να προβούν στι απαραίτητε μεταρρυθμίσει ακολουθώντα του κανόνε που έχουν αποφασιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Τώρα ο κύριο Ντότ. Δεν είναι εδώ. Δίνω αμέσω το λόγο στον κύριο Μισελ Νταντά. Έχει, έχει το λόγο. Κύριε Επίτροπε, λέτε ότι η μελλοντική σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας επιτρέπει στην ΠΑΚ να έχει δίκτυα ασφαλείας μέσα από σύγχρονους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς. Οι παρελθούσες κρίσεις επέδειξαν τις αδυναμίες και τις ΚΑΠ και των αγορών. Μιλήσατε εσείς για τα μέσα που θα χρησιμοποιήσετε προηγουμένως. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα πράγματα όμως για αυτά τα μέσα. Και πώς βλέπετε εσείς ως μέσο την σύναψη συμβάσεων ανά γεωργικό κλάδο ή αναπροϊόν. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εμποδίσει τον ανταγωνισμό ή όχι. Για τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς, εγώ μιλάω για σύγχρονους μηχανισμούς που δεν θα διακυδεύουν την λειτουργία της αγοράς. Αναφέρομαι εδώ σε μερικούς ειδικού μηχανισμούς, ας πούμε ε, εγγυητικά ταμεία, ε, ασφαλίσεις για την εγγύηση των εισοδημάτων, όταν δηλαδή πλήττονται ουσιαστικά τα γεωργικά εισοδήματα για τα οπορολαχανικά θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους μηχανισμούς και να τους διευρύνουμε και σε άλλους τομείς. Μιλήσατε τώρα για τη σύμβαση, για τη μεθόδο της σύναψης συμβάσεων. Εμείς πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει και αυτό το σύστημα, να μπορέσουμε εμείς μέσα στα πλαίσια των διαφόρων δικτύων να δώσουμε κίνητρα στους γεωργούς ε, χωρίς να στρεβλώσουμε τους κανόνες του ανταγωνισμού. Εγώ θα ήθελα να παροτρύνω τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή να δώσουν ορισμένες δυνατότητες παρεκκλήσεων για ορισμένα προϊόντα λαμβάνοντας υπόψη και τον ιδιάζοντα χαρακτήρα της γεωργίας για να μπορέσουμε να φέρουμε σε ισορροπία την προσφορά με τη ζήτηση, να μπορέσουν οι αγορές να λειτουργήσουν καλύτερα. Δεν θα πούμε πώς θα λειτουργήσουν οι αγορές, αλλά θα τις βοηθήσουμε να λειτουργήσουν καλύτερα. Ένα ταμείο εγγύσεων για τη διασφάλιση του εισοδήματος των γεωργών και εδώ μπορεί να υπάρξει ε, υπογραφή ε, συμβάσεων Εμείς έχουμε μερικούς μηχανισμούς από το παρελθόν που θα μπορούσαμε να προσαρμόσουμε. Αλλά και οι άμεσες πληρωμές και αυτές μπορούν να διασφαλίσουν τη σταθερότητα των εισοδημάτων των γεωργών. Τώρα η ισορροπία προσφοράς και ζήτησης επίσης. Στα παλιά μέσα που είχαμε στη διάθεσή μας είχαμε τη ρύθμιση της παραγωγής. Εσείς μιλήσατε για το πόσο υποστηρίζεται τα προϊόντα ποιότητας. Αυτά τα προϊόντα όμως μπορούν να χρησιμοποιήσουν... Μπορούμε λοιπόν εμείς να χρησιμοποιήσουμε αυτό το παλιό εργαλείο, διότι ξέρετε η ποιότητα δεν είναι το παν. Η τιμή απαιτεί μια ρύθμιση της ποσότητας στην αγορά. Μα εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα ε, βασικής λειτουργίας της αγοράς. Μιλήσατε εσείς ε, για ποιότητα, για προϊόντα προέλευσης, ε, γεωγραφική προέλευση κλπ. Πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι καλύτεροι μηχανισμοί που διασφαλίζουν τη συνέχεια και την ισορροπία σε επίπεδο παραγωγής για να μην αποδυναμωθεί ένα προϊόν με ειδικά χαρακτηριστικά ποιότητας στην αγορά. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία συνδέονται διάρκεια με την αγορά και θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να το σκεφτούμε. Πρέπει να δούμε εμεί πώς θα τα διαχειριστούμε όλα αυτά στο μέλλον. Ο κύριος Ταμπατζή. Πες μου, κύριε Τσόλο, πώς ε, θα ρυθμιστεί αυτή η αστάθεια και η εναλλακτικότητα, η τάση αλλαγής των γεωργικών αγορών. Πώς ε, θα οικοδομήσουμε εμείς αυτές τις νέες αγορές και θα τις ρυθμίσουμε όταν η, η δημόσια παρουσία έχει εξαφανιστεί από τη γεωργία, πώς θα ενισχύσουμε εμείς τους παραγωγούς όταν τα σούπερ μάρκετ ελέγχουν τα πάντα, όταν τα μεγάλα δίκτυα διανομής ελέγχουν τα πάντα στη γεωργία. Κουράγιο, κουράγιο λοιπόν. Μα σχετικά με αυτήν την ε, συνεχή αλλαγή της γεωργίας. Ε, ε, εγώ μιλάω, όπως επίσης και την εποχικότητα της γεωργίας, και όταν υπάρχει μια μεγάλη διακύμανση μιλάω για τη δημιουργία να ας πούμε αυτού του ταμείου ασφαλίσεων που θα εγγυάται το εισόδημα των γεωργών. Τώρα έλεγα συμβάσεις και το συνδέω εδώ και με το δεύτερο ερώτημα για τα σούπερ μάρκετ και τη μεγάλη διανομή. Μα και αυτό μπορεί να ρυθμιστεί με διαπραγματεύσεις για τον τρόπο με τον οποίο η προστιθέμενη αξία κατανέμεται μέσα στην, στο όλο δίκτυο. Το κάνουμε, αρχίσαμε δηλαδή να το κάνουμε για τα γαλακτοκομικά μπορούμε να το κάνουμε και για τους άλλους τομείς. Αλλά εδώ δεν μιλάω για δημόσια παρέμβαση. Οι αγορές πρέπει να λειτουργήσουν και η ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης να ορίζει τα πράγματα. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια διαπραγμάτευση μέσα στα ίδια τα δίκτυα και θα πρέπει να ενισχύσουμε τους ίδιους τους γεωργούς ούτως ώστε να συνεταιρίζονται και να μπορούν να συμμετέχουν πιο δυναμικά στις διαπραγματεύσεις. Άμα δείτε εσείς ε, την ε, κατανομή της προστιθέμενης αξίας θα δείτε ότι πολλές φορές το περιθώριο κέρδους δεν είναι μόνο η μεγάλη διανομή που το κερδίζει γιατί υπάρχουν και άλλοι μεσάζονται στη μέση. Ευχαριστώ. Μάριαν Χάρκιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, στην παρουσίασή σας σήμερα το πρωί είπατε ότι η ΚΑΠ θα πρέπει να διασφαλίσει καταρχάς το σωστό εισόδημα και την επιστηστική ασφάλεια. Φυσικά αυτά τα δύο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, γιατί αν δεν έχουν σωστό εισόδημα οι αγρότες δεν θα έχουμε ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι ένα από τα θέματα που προκαλεί, ε, αν θέλετε, μη θεμητά εισοδήματα στους αγρότες είναι η πίεση στην αγορά και πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο δημιουργήθηκε μια υπηρεσία για να εξεταστεί στο ελεύθερο εμπόριο η τήρηση κάποιων δεντολογικών αρχών. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τις απόψεις σας για το θέμα αυτό. Τι μέτρα θα λάβετε, αν λάβετε μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι θα υπάρχει ισορροπία μεταξύ των ε, παραγωγών και των μεταποιητών. Να υπάρξει δηλαδή μια διόρθωση αυτή της ανισορροπίας ε, απάντηση. Όπως στη Ρουμανία όταν ήμουν υπουργό ε, Αγροτικών Υποθέσεων, παρότρινα τους παραγωγού και τους μεταποιητέ να προβαίνουν σε διαπραγματεύσεις και είχαμε τέτοιου είδους πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές αλλά νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει μεταξύ των φορέων των ίδιων στην τροφική αλυσίδα. Ως Επίτροπος μπορώ να ενθαρρύνω τέτοιου είδους συζητήσεις. Δεν νομίζω όμως ότι την παρούσα φάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρέμβει στη σχέση μεταξύ των παραγωγών και των μεταποιητών των ελληνεμπόρων. Νομίζω ότι αυτός ο κώδικας ε, δεντολογίας ε, για τις σχέσεις αυτές θα μπορούσε να αποτελέσει μία λύση. Αλλά θα πρέπει πρώτα να υπάρχει μία συμφωνία και των δύο μερών. Γενικά όμως, όπως είπα και στην, ε, στον κ. Ταμπατζή, θεωρώ ότι μεταξύ των διαφόρων φορέων οι επαφές αυτές θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε καλύτερη ρυθμιστική κατανομή και να προσθέσουν αξία στην τροφική αλυσίδα. Ως Επίτροπος, λοιπόν, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ενθαρρύνω, να παρατρύνω τέτοιου είδους συζητήσεις, γιατί πρόκειται για ένα θέμα το οποίο σχετίζεται και με τον ανταγωνισμό. Επερώτηση. Ναι, ευχαριστώ υποψήφια επιτρόπε, καταλαβαίνω λοιπόν τι λέτε, αλλά ήλπιζα με κάποιο τρόπο η ομάδα υψηλού επίπεδου για τον ε, ανταγωνιστικότητα του αγροτοφικού κλάδου θα μπορούσε να παρέμβει κατά κάποιο τρόπο για να προωθήσει το θέμα αυτό. Καταλαβαίνω τι λέτε φυσικά, ότι το μόνο που μπορείτε να κάνετε εσείς ουσιαστικά είναι να δώσετε κίνητρα, να ενθαρρύνετε τους φορείς για να εργαστούν κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο, αλλά θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό με την ομάδα υψηλού επίπεδου, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο ε, στρεβλώνει τις, αγο... τις τιμές και πραγματικά προκαλεί προβλήματα. απάντηση. Κατά τους επόμενους μήνες θα παρουσιάσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα συμπεράσματα των πορίσματα των συζητήσεων της ομάδας ε, υψηλού επίπεδου και είμαι αισιόδοξο ότι θα υπάρξουν καλά αποτελέσματα προκειμένου να αναλυθεί η δυνατότητα να δοθεί συνέχεια στα αποτελέσματα αυτά και στα, στις μεθόδους αυτές ε, και σε άλλους κλάδους. Όλα αυτά σας συνεργασία με τους συναδέλφους από τον ανταγωνισμό, γιατί θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφορετικών κλάδων για να υπάρχει κάποια απόκληση από τους κανόνες ανταγωνισμού, γιατί επειδή είναι κοινή η αγορά θα πρέπει να υπάρχουν και κοινοί κανόνες. Αλλά είμαι έτοιμος να εξετάσω όλες τις ε, λύσεις που έχουμε στη διάθεσή μας για να ενισχύσουμε τους ε, παραγωγούς και σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για την τροφική αλυσίδα. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος και τώρα περνάμε στον κύριο Μποβέ. Oui, ε, Ο Ζωζέ, για ένα πιο... Σφαιρικό θέμα. Λοιπόν, εξαρτόμαστε από ορυκτές πηγές ενέργειας. Δύο τόνοι ανακάτοικο πετρέλαιο καταναλώνει η Ευρώπη. Και αυτή η κατανάλωση στον αγροτικό τομέα του πετρελαίου είναι υπεύθυνη για το 2% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος. Μέχρι τώρα η γεωργική πολιτική της Ένωσης τι έκανε. Αύξησε την καταστροφή για παράδειγμα, εντατικές καλλιέργειες καλαμποκιού οδήγησαν σε διάβρωση του εδάφους ή αποψήλωση ή εγκατάλειψη των γεών και τα λοιπά οδήγησαν στην διάβρωση των εδαφών. Τι θα κάνει η Κομισιόν όμως για να ενισχύσει το σχέδιο των νέων αγροτών που θέλουν να διορθώσουν όλα αυτά τα κακό σκήμενα. Το είπα. Τα θέματα της ε, κλιματικής αλλαγής και η προστασία του περιβάλλοντος συμβαδίζουν με την γεωργία μας. και την πολιτική μας για τη διαμόρφωση του υπεύθυνου καταναλωτή. Εμείς θα, τα πρέπει, θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε και περιφερειακά, να δούμε τι χρειάζεται στη μία περιοχή, τι χρειάζεται στην άλλη και θα το δούμε και με τη συνάδελφο για την έρευνα. Να δούμε τι είδους έρευνα μπορούμε εμείς να εφαρμόσουμε, τι ειδικαικούς μηχανισμούς για την ενίσχυση του Γιωργού για προς την καινοτομία. Η αξιολόγηση δε της τοπικής γεωργίας και αυτό μπορεί να βοηθήσει. Μέχρι τώρα εμείς επιμείναμε πολύ στην βιομηχανική γεωργία. Σήμερα και η τοπική γεωργία μπορεί να ενισχυθεί σε ορισμένες περιοχές προς τον τόπιο καταναλωτή και να πούμε ότι αυτές οι τοπικές αγορές είναι κομμάτι των κοινοτικών αγορών. Και φυσικά αυτός είναι ένας τρόπος για να ενθαρρύνουμε αυτή την πιο, τη γεωργία που θα σέβεται περισσότερο και τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. Ο Ζωζέ. Παράρτημα. Επερώτημα, συγγνώμη. Που αφορά στο εισόδημα των γεωργών. Κάτι δεν άκουσα ακόμα από εσά. Η Ευρώπη στα πλαίσια του ανταγωνισμού απαγορεύει στην, στα σούπερ μάρκετ να πολλούν με απώλεια. Γιατί τόσο στα οπόρα λαχανικά όσο και στα στο γάλα και σε άλλα προϊόντα πρέπει εμείς να έχουμε κρίσεις γιατί τι, Διότι οι γεωργοί πουλούν με χασούρα. Και ο Ρούσβελτ αυτό το είχε νομοθετήσει. Απαγορεύοντας τους γεωργούς να, πληρούν, να πουλούν τα γεωργικά τους προϊόντα με χάσιμο. Μα κοιτάστε εδώ είναι λεπτό το ερώτημα. Διότι ένας έμπορος αγοράζει ένα προϊόν σε μια αλφα τιμή και το πουλάει σε β τιμή. Και μπορεί να κάνει και έκπτωση να το πουλήσει λιγότερο από όσο το αγόρασε. Τώρα, για το Γιωργό πολλές φορές πουλάει με χασούρα αντισταθμίζοντας αυτό το οποίο ε, κέρδισε την προηγούμενη χρονιά. Πρέπει να βρεθεί όμως ένας μηχανισμός ούτως ώστε ο Γιωργός να μην υποχρεούται να πληρώνει, να πουλάει συγγνώμη με απώλεια το προϊόν του. Πρέπει όμως εμείς να βοηθήσουμε και τον Γιωργό να αποκτήσει ανταγωνιστικότητα έναντι της ε, τιμής που του προσφέρουν. Δεν ξέρω τι περιθώρια μπορώ να έχω εγώ ως ε, Επίτροπος για τη Γεωργία για να εξετάσω αυτό το ζήτημα. Να δούμε από πού προέρχεται αυτή η χασούρα για τον Γιώργο. και ε, για να μπορέσω δηλαδή να βρούμε και τη λύση ώστε να μην χρειάζεται να ξεπουλάει ο Γιώργος για να ζήσει. Ο κύριος Βοσεβός, κύριε, ευχαριστώ. Κύριε υποψήφι. επίτροπε, είμαι ευτυχής που μπορώ να θέσω ένα ερώτημα προς έναν υποψήφιο επίτροπο από νέο κράτος μέλος, γιατί έχει να κάνει το θέμα αυτό και με διακριτική μεταχείριση σε ό,τι αφορά τι επιδοτήσει. Η προηγούμενη Επιτροπή πρότεινε την εξή λύση. Μετά το 2013 το επίπεδο των επιδοτήσεων να προβλέψει κάποιες χώρες με διακριτική μεταχείριση και κάποιες άλλες με προνομιακή μεταχείριση. Από αυτές που θα υποστούν διακριτική ε, μεταχείριση είναι και κάποιες καινούριες και κάποιες μικρές, ε, κάποιες μεγα... και κάποιες και παλιές ε, χώρες και υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην διαδικασία αποδέσμευσης. Τι σκοπεύετε να κάνετε λοιπόν για να μην υπάρχει τέτοια διακριτική μεταχείριση κατά τόσο μεγάλο αριθμό κρατών μελών. Απάντηση. Όπως είπατε αξιότιμα κύριε Βουσκευσκή, το θέμα του κριτηρίου για την εκχώρηση των άμεσων ενισχύσεων θα το πρέπει να συζητήσουμε και μάλιστα πριν από τις προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Και αυτό θα αποτελέσει μία ευκαιρία να διαμορφώσουμε λύσεις και με την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τις οποίες τελικά θα καταφέρουμε μεγαλύτερη ισορροπία. Οι διαφορές αυτές ε, δικαιολογούνται από κάποια άποψη λόγω των διαφορετικών όρων, συνθήκων που επικρατούν για την γεωργική παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, στόχος θα πρέπει να είναι να υπάρχουν σαφή και διαφανή κριτήρια με τα οποία θα αποφύγουμε τέτοιες διακριτικές μεταχειρήσεις και τους επόμενους μήνες όταν θα συζητήσουμε το μέλλον της ΚΑΠ θα βρούμε από κοινού λύσεις για το ποια κριτήρια θα πρέπει να εφαρμοστούν όταν θα καταργηθούν τα ιστορικά κριτήρια. Σας ευχαριστώ, Επίτροπε, για την απάντηση αυτή. Θα ήθελα να πω το εξή. Τα θέματα αυτά σχετίζονται και με τον προπολογισμό, αλλά το θέμα δεν είναι να πάρουμε χρήματα από αυτούς που έχουν πιο πολλά χρήματα και να τα δώσουμε σε άλλους. Όχι. Το θέμα είναι να δώσουμε πιο πολλά σε αυτούς που τα χρειάζονται. Χαίρομαι λοιπόν που θα προασπιστείτε τον προπολογισμό του ΚΑΠΑ αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι μεγαλύτερο προπολογισμό για την ΚΑΠΑ, γιατί μετά την Λισαβόνα θα υπάρξει περαιτέρω ευρωπαϊκή ενοποίηση, άρα θα πρέπει να έχουμε και πιο πολλά κονδύλια. Και νομίζω ότι η γεωργία αποτελεί ένα από τα βασικά μας ε, θέματα για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Θα είσαστε υπέρ μιας προσέγγισης όπου κάθε χώρα θα ρυθμίζει αξεχωριστά το καθεστώς που θα ισχύει σχετικά με τους γενετικά τραποποιημένους οργανισμούς. Απάντηση. Ναι. Έχει υποβάλει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήδη μια τέτοια προσέγγιση και την οποία και υποστηρίζω επί της αρχής. Οι επιστημονικές μελέτες, τα επιστημονικά πορίσματα από τη στιγμή που αποφανθούν ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι για τον καταναλωτή, για την υγεία του καταναλωτή και για το περιβάλλον από τα προϊόντα αυτά, από τη στιγμή λοιπόν που αυτό θα καταδείξουν τα επιστημονικά απορίσματα, δεν υπάρχει κάποιος λόγος και θα μπορέσουν οι ρυθμίσεις αυτές να λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, γιατί υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις και στάσεις. Αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Υπεύθυνο και αρμόδιος είναι ο συνάδελφός μου για θέματα προστασίας του καταναλωτή και υγείας. Μάλιστα και τώρα περνάμε στον κύριο Μέσσερ Σμιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι από την Δανία, όπου έχει συμφωνηθεί από όλα τα κόμματα ότι η ενίσχυση των αγροτικών ε, προϊόντων ε, βλάπτει τους παραγωγούς, τους καταναλωτές και την Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν διαπιστώνουμε ότι η γραμμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της κυρίας Φισερμπέλ τα τελευταία χρόνια ήταν ακριβώς αυτή για την κατάργηση των ενισχύσεων. Ακούσαμε πρόσφατα έναν συνάδελφο, τον κύριο Λεβαντόφσκι, ο οποίος είπε ότι τα επόμενα πέντε χρόνια δεν θα συνεχιστεί αυτή η γραμμή. Μίλησε ο Λεβαντόφσκι για την κατάργηση της σταδιακής ε, αναστολής, κατάργησης των επιδοτήσεων. Δεν θέλουμε δηλαδή να μειωθούν οι επιδοτήσεις, αλλά να αυξηθούν ή να μείνουν στο παρόν επίπεδο. Εσείς, σύμφωνα με τον κύριο Λεβαντόφσκι, ή θέλετε ότι θα πρέπει να καταργηθούν σιγά σιγά οι επιδοτήσεις, ο Επιτροπός. Δεν γνωρίζω, δεν ξέρω αν η Μαριάν Φίσερ Μπέλ είχε θέσει στόχο να μειώσει τις επιδοτήσεις, αλλά θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ισορροπία μεταξύ των άμεσων επιδοτήσεων του πρώτου πυλώνα και της ε, ανάπτυξης της υπαίθρου στο δεύτερο πυλώνα. Εισήχθη αυτός ο μηχανισμός για να ενισχυθεί η ε, ανάπτυξη της υπαίθρου, ο δεύτερος πυλώνας και το θέμα αυτό δεν τίθεται πλέον, γιατί στην ΚΑΠ μετά το 2013 μαζί με τα κράτη-μέλη θα έχουμε τη δυνατότητα να αποφασίσουμε από κοινού. Ποιος, ποιο κομμάτι του προπολογισμού θα μείνει στον πρώτο πυλώνα και ποιο θα μεταφερθεί στο δεύτερο πυλώνα. Και όπως σας είπα, αυτές οι επιδοτήσεις και οι άμεσες ενισχύσεις έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν για την σταθερότητα των εισοδημάτων και των αγροτών στην Δανία. Και είναι σημαντικό αυτό ο μηχανισμό. Θα πρέπει να διατηρηθεί. Αλλά πρέπει να υπάρχει η ισορροπία μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα. Και έχουμε την ευκαιρία να προβούμε σε εκ νέου, αν θέλετε, διαμόρφωση της ισορροπίας αυτής στις συζητήσεις για την ΚΑΠ μετά το 2013. Αλλά είναι σημαντικός ο ρόλος τους και όπως σας είπα θα πρέπει να διασφαλίσουμε ένα ελάχιστο εισόδημα για τους γεωργούς και νομίζω ότι θα πρέπει να παραμένουν οι υπεδοτήσεις. Επερώτηση. Ο κύριος Λεβαντόφσκι τάχθηκε υπέρ μάλλον ακούστηκε Μα ο κ. Λεβαντόφς και ανοιχτά υπέρ της συνέχισης των επιδοτήσεων. Σας ερωτώ συγκεκριμένα, συμφωνείτε ότι θα πρέπει να μειωθούν οι επιδοτήσεις για να φτάσουν σε ποσοστό 40% γιατί πολλοί στη χώρα μου δεν είναι ευχαριστημένοι όταν δαπανάτε τέτοιο μεγάλο ποσό και θεωρούν ότι θα πρέπει να μειωθεί οι επιδοτήσεις. Να μην εξαρτάται δηλαδή η γεωργία από τον κρατικό κορβανά. Γι' αυτό λοιπόν ρωτώ, θα ταχθείτε υπέρ της μείωσης βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα των επιδοτήσεων. Απάντηση. Νομίζω ότι κάπου χρειάζεται ένα συνεκτικό προϋπολογισμό. Δεν μιλάμε μόνο για τα κονδύλια τα οποία ωφελούν μόνο τους παραγωγούς. Όχι, μιλάμε για τα τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για τον αγροτροφικό κλάδο, ο οποίος δεν είναι σημαντικός μόνο για την ενιαία αγορά, για τις θέσεις εργασίας και τις εμπορικές σχέσεις, αλλά έχει και μια επιπλέον σημασία. Το είπαμε ήδη ότι ο προπολογισμό αυτός έχει βάσεις, είναι δικαιολογημένος επειδή έτσι διασφαλίζουμε την παραγωγή για την Ευρώπη και δεν ε, επιτρέπονται σφάλματα να επιτρέψουμε να μειωθεί η παραγωγή, γιατί τότε θα αυξηθεί το κόστος. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό θεωρώ ότι ο, υψηλο, υψηλός προϋπολογισμός για την γεωργία είναι απόλυτα δικαιολογημένος. Έχουμε τα σχετικά επιχειρήματα, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την μεταρρύθμιση, την αναθεώρηση, για να το καταστήσουμε γνωστό αυτό, να εξηγήσουμε γιατί είναι τόσο σημαντική η στήριξη της παραγωγής και θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι σωστός, να παραμείνει σωστός ο εμπεριπολογισμός για τη γεωργία. Θα πρέπει να ζητήσουμε τρόπους για να γίνει καλύτερη κατανομή μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα χωρί να δοθεί σε κίνδυνο το εισόδημα το αγροτικό. Ωραία, προχωράμε στο τέταρτο γύρο. Είμαστε ακριβώ στην ώρα μα. Έχουμε και ένα λεπτό από του σοσιαλιστέ λόγω τη εξοικονόμηση χρόνου του συναδέλφου Ταμπάζη. Πάμε λοιπόν ε, γρήγορα γρήγορα για να δώσουμε χρόνο και σε άλλους συναδέλφους. Ο κύριος Σεγκερέσκι τώρα. Ο προηγούμενος ομιλητής είπε ότι χάνουμε μεγάλα ποσά για, από διάφορες πολιτικές. Η Γεωργία, όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θεωρούν ότι είναι σταθεροποιημένη η κατάστασή τους. Δεύτερο πρόβλημα, μιλήσατε για σύγχρονους μηχανισμούς της αγοράς. Μπορείτε αυτό να μου το εξηγήσετε. οι πληρωμέ θα πρέπει να βασίζονται στην επιφάνεια ή απλά στην δραστηριότητα, ανάλογα με το αν η επιχείρηση είναι ενεργή. Σε πολλά κρατημέλη υπάρχει μεγάλο κατακαιρματισμό των γεωργικών επιχειρήσεων με μια άλλη συνδυασμό, με άλλη δραστηριότητα. Ποιοι Ποιου προσανατολισμού στήριξη προβλέπετε εσεί για τέτοιου είδου γεωργικέ δραστηριότητε, Ποια είναι η θέση αυτών των ε, γεωργικών επιχειρήσεων στην αγορά και έπειτα δεν θα γίνει μεγαλύτερη διαδικασία συγκέντρωσης των γεωργικών επιφανειών. Ευχαριστώ. Δεν αισθάνονται όλοι οι γεωργοί την σταθερότητα που προσφέρει ΚΑΠ. Υπάρχουν ορισμένες περιοχές ε, συμπεριλαμβανομένης και της δικής σας χώρα, όπου στο μέλλον το επίπεδο των άμεσων πληρωμών θα αυξηθεί γιατί η χώρα σας ξεκίνησε από ένα χαμηλότερο επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνει και άλλη μια προσπάθεια, δηλαδή αναδιάρθρωση και εξυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων. Και από αυτή την άποψη η κοινή γεωργική πολιτική θα ε, λειτουργήσει με τους μηχανισμούς της. Ε, τώρα όσον αφορά τους σύγχρονους μηχανισμούς της αγοράς, το έχω ήδη πει, δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες, γιατί πρόκειται εδώ για τεχνικά στοιχεία τα οποία πρέπει να ορίσουμε με τους ε, ειδικού. Πιστεύω ωστόσο ότι η δημιουργία Ταμείου Εγγύσεων, για παράδειγμα, που να μπορεί να εξασφαλίσει τη σταθερότητα των εισοδημάτων των γεωργών ή τις παρεμβάσεις στη στιγμή που μειώνεται το εισόδημα των γεωργών με πολύ δραματικό τρόπο. Φυσικά, σε ορισμένου γεωργικού τομεί η κατάσταση θα είναι διαφορετική. Η δημιουργία ενό τέτοιου ταμείου θα μπορούσε να αποτελεί μια λύση, κατά την άποψή μου. Ταυτόχρονα, ανα τομέα, ορισμένα είδη συμβάσεων θα μπορούσαν να διασφαλίσουν αυτή τη σταθερότητα τιμών αλλά και εισοδημάτων των γεωργών. Θα δούμε αν θα μπορέσουμε να βρούμε και άλλες λύσεις. Αλλά κατά την άποψή μου το γεγονός ότι υπάρχουν αυτές οι ανησυχίες και ότι τις συζητάμε αποτελούν ήδη ένα καλό σημείο κίνηση όσον αφορά τις μικρές εκμεταλλεύσεις, ε, τις ε, οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Ο τρόπος με τον οποίο ε, βοηθούνται οι πληρωμές ανά εκτάριο δηλαδή θα ε, ευνοήσει την κατάσταση. Όμω μέσω του δεύτερου πυλώνα τη κοινή γεωργική πολιτική μπορούμε να βρούμε σε ορισμένε περιοχέ και κατηγορίες ε, ε, γεωργών μπορούμε να εντοπίσουμε μηχανισμού συγκεκριμένου που να είναι καλύτερα προσαρμοσμένοι. Τώρα, για την απασχόληση και για τον τρόπο με τον οποίο η γεωργία δημιουργεί ή διατηρεί τις θέσεις απασχόλησης. Αυτή είναι μια ιδέα η διατηρει τι θεσει απασχοληση αυτη ειναι μια ιδεα η οποια μου είναι ιδιαίτερα προσφυλή. Θα πρέπει να βρούμε ένα συγκεκριμένο μηχανισμό για, δείκτες μέσω των οποίων θα μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Γνωρίζω ότι μέσα στο πλαίσιο, μέσα στις υπηρεσίες της Κομισιόν υπήρξε μια τάση παλιότερα να ε, δεχτούμε τέτοιου είδους ε, νέους δείκτες, αλλά για την ώρα δεν έχουμε, βρει, δεν έχουμε καταλήξει στο πώς θα αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο των μέτρων. Σικέρσκι. μιλάτε για εξυγχρονισμό μεταρρύθμιση. Όλα αυτά κοστίζουν όμως. Πού θα βρούμε τα χρήματα για να πληρώσουμε τον εξυγχρονισμό και έπειτα πώς θα μπορέσουμε να εγγυηθούμε ένα ενιαίο σύστημα άμεσων πληρωμών διατηρώντας την απέτηση της στήριξης για τους γεωργούς που, δουλεύουν σε δυσμενείς ζώνες όπου ε, επικρατούν μεγάλες ε, δυσκολίες και έπειτα μπορείτε να δώσετε τη δυνατότητα στήριξης για πολύ συγκεκριμένες παραγωγές όπως ε, τα καπνά που είναι χαρακτηριστικό για χώρες όπως η Πολωνία, η Ιταλία και η Ελλάδα και μάλιστα με τις μικρές εκμεταλλεύσεις που καλλιεργούν καπνά. Οι νέε πληρωμέ μέσω των νέων ρυθμίσεων για τη νέα ΚΑΠΑ θα διασφαλίσουν την μεγαλύτερη ισότητα. Αυτό το έχω πει, το έχω υπογραμμίσει. Είναι μία από τις προτεραιότητές μου και ένα από τα στοιχεία προσαρμογής του πρώτου πυλώνα. Και ελπίζω πως σε αυτή την κατάσταση θα βρίσκονται και οι γεωργοί για τους οποίους κάνατε λόγο σε σχέση με την ισότητα. Βεβαίως εκεί όπου ορισμένε παραγωγές δεν είναι αποδοτικές μέσω του δεύτερου πυλώνα της ΚΑΠ, μέσω των επενδύσεων στον εξυγχρονισμό υπάρχει δυνατότητα για τους γεωργούς να στραφούν σε παραγωγές πιο αποδοτικές, αλλά βεβαίως θα λαμβάνουν, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ζήτηση στην αγορά. Ε, όσον αφορά την παραγωγή καπνού, ξέρετε ότι ήδη υπάρχει μία απόφαση, έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και ανάλογα με το περιθώριο ελιγμού που έχουν τα κράτη-μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 68 για την καταβολή των άμεσων πληρωμών, μπορούμε να βρούμε μεταβατικές λύσεις και για αυτό το τομέα. Ωραία. Τώρα ο κύριος Μάρκα Ταραμπέλα. Κύριε υποψήφιο επίτροπε, με μεγάλη λύπη μοιράστηκα το 2009 με τους γαλακτοπαραγωγούς που οδηγήθηκαν να πετάξουν την παραγωγή τους γιατί δεν ε, ε, πληρώνονταν αρκετά. Και αυτό οφείλεται στην απορρίθμιση των αγορών για την οποία μιλάμε. Λύπη και θλίψη για τροποποίηση και ρύθμιση σύγχρονη συμβάσεις στους ε, διαφόρους κλάδους και στρέφουμε τα νότα μας σε πιο αποτελεσματικές λύσεις Επίσης, η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη στρέφουν τα νότα τους στις ποσοστώσεις που επέτρεψαν να λειτουργήσει κάπου εδώ και 15 χρόνια, ε, εδώ και 25 χρόνια και μήπως θα έπρεπε αναμένοντας αυτού τους νέους κανόνες ε, θα εγκαταλείψετε τελείως τις ποσοστώσεις, θα προσπαθήσετε να πείσετε τα κράτη-μέλη και τους συναδέλφους των Επιτροπ... της Επιτροπής να συνεχίσουν να τα χρησιμοποιούν. Και θα μιλήσω και για τη ζάχαρη στην επερώτηση, άλλη απορρίθμιση και σχέση με τις αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις. Επίσης θα εγκαταλείψετε τελείως τις αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις που επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να βοηθήσουν τις πιο ειστερούσες ε, ε, ε, περιοχές. Τώρα για τις ποσοστώσεις δεν το εγκαταλείπω εγώ. Είναι μια συζήτηση που έχει γίνει στο Συμβόλαιο μαζί με τα κατημέλη και έχει ληφθεί σχετική απόφαση. Πιστεύω ότι το να επανερχόμαστε σε ένα τέτοιο μηχανισμό και μπορεί να αποσταθεροποιήσει ακόμα και τους γεωργούς και τις αγορές γιατί έχουμε μια απόφαση, έχουμε, μια, έχουμε μάλλον ξεκινήσει σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και η λύση δεν είναι να στρεφόμαστε νοσταλγικά προς το παρελθόν, αλλά βρούμε τρόπους με τον οποίο ο περιορισμός των ποσοστώσεων που ανοίγει ευκαιρίες για ορισμένες ε, κτηνοτρόφους να μην επηρεάσει συγκεκριμένες περιοχές όπου υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα. Τώρα, για τις ιδιαίτερες περιοχές με τις ειδικά προβλήματα στο γαλακτοκομικό τομέα θα πρέπει να βρεθούν και τα κατάλληλα και προσαρμοσμένα μέσα. Με αυτό εγώ θα ασχοληθώ, αλλά δεν πιστεύω πως ε, στις συνθήκες τις οποίες δουλεύουμε και ανοίγουμε τις αγορές μας ε, Τη ευρωπαϊκή η συντήρηση των ποσοστώσεων θα ήταν λύση, γιατί οι ποσοστώσει ανταποκρίνονται ίσω σε ένα πρόβλημα μεταβλητότητα τη προσφορά, αλλά όχι τη ζήτηση και η κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε πρόσφατα με τη μείωση τη ζήτηση, ακόμα και με τη συντήρηση, τη διατήρηση μάλλον των ποσοστώσεων, δεν μπορούσαμε να έχουμε ρυθμίσει το πρόβλημα. Και γι' αυτό και πιστεύω πω ε, ποσοστα... οι ποσοστώσει δεν είναι ο κατάλληλο μηχανισμό. Αλλά αυτό δεν μα εμποδίζει να βρούμε μηχανισμού που να μα οδηγήσουν σε κάποια σταθερότητα στον γαλακτοκομικό τομέα, ιδιαίτερα στι λιγότερο ευνοούμενε ε, περιοχέ ε, και που εξαρτώνται εν μέρη από τη γαλακτοκομική παραγωγή. Ήδη στο απολογισμό υγεία μπορέσαμε να, δούμε, ε, να βρούμε αυτή τη λύση με το άρθρο 68 που μας επιτρέπει να παρεμβαίνουμε με ιδιωτικό τρόπο. Πιστεύω πως αυτά τα ειδικά στοιχεία θα πρέπει να τα δούμε και στη συνέχεια γιατί από ό,τι κατάλαβα υπάρχει ανάγκη για κατάλληλες λύσεις για ορισμένες περιοχές. Ευχαριστώ, Επίτροπο. Ήθελα, όπως σας το είπα, να σας μιλήσω μετά από το γάλα για τη ζάχαρη. Η ΚΟΑ υπέστη κάποιες ε, τροποποιήσεις εδώ και κάποιε χρόνια και μέχρι σήμερα η παραγωγή ήταν ε, ε, υπερβολική. Έχουμε δηλαδή πλονάσματα, αλλά μπορούμε να εξάγουμε μόνο 1.350.000 τόνους, ενώ η παγκόσμια αγορά ζητά σήμερα 7 εκατομμύρια τόνους. Είναι ελληματική η παγκόσμια αγορά και ενώ η διεθνής ε, τιμή αυξάνεται, η ευρωπαϊκή τιμή είναι στα 400 περίπου ευρώ, θα μπορούσαμε να εξάγουμε χωρίς καμία δημόσια παρέμβαση, ούτε επιστροφή και παρεμποδιζόμαστε. Είναι μια απορρίθμιση, μια μη λειτουργικότητα της αγοράς, την οποία αναφέρατε στη αρχική σας ε, παρέμβαση. Είναι ένα, μια αποτυχία της αγοράς και αν πια γίνεται επίτροπε στις 27 Ιανουαρίου το πρωί, θα παρέμβετε για αυτό το ζήτημα. Και αν ναι, με ποιο τρόπο. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα περιθώρια λιγμού ε, που μας δίνει η μεταρρύθμιση που αποφάσισαν τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο και σε σχέση με τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην ε, διεθνή αγορά. Είναι ένα θέμα όμως που αν με βεβαιώσετε τις 27 θα ασχοληθώ πιο συγκεκριμένα για να μπορέσω να σας δώσω μια απάντηση γιατί νομίζω πως αυτό αξίζει να μελετηθεί με λεπτομέρειες για να δούμε ακριβώς το περιθώριο λιγμού για τη μεταρρύθμιση που έχουμε ήδη αποφασίσει, αλλά και το περιθώριο λιγμού που μας επιτρέπουν οι διεθνείς συμφωνίες. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω περισσότερο, γιατί χρειάζομαι τις λεπτομέρειες. Ωραία. Επίτροπε, τώρα είναι η σειρά της Ελίζαμπετ Κόστιγκερ. Κυρία Τσόλος, είπατε στην αρχή ότι οι περιοχές με φυσικές, ε, φυσιονικά μειονεκτήματα, ιδιαίτερα για ορεινές περιοχές, θέλετε να συνεχίσουν να λαμβάνουν ενίσχυση. Μπορείτε να εγγυηθείτε την επαρκή οικονομική ενίσχυση και πώς θέλετε να εκπροσωπήσετε τα συμφέροντα αυτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα ήθελα να ακούσω σε ό,τι αφορά τις ορεινές περιοχές αν θα συνεχίσετε το έργο των τελευταίων ετών ή αν θα χαράξετε νέους δρόμους. Ο Επίτροπος. κοιτώντας, ε, μάλλον αν εξοπλίσουμε σωστά τον δεύτερο πυλώνα, στην επόμενη συζήτηση για την ΚΑΠ μετά το 2013, δηλαδή τους επόμενους μήνες, τον επόμενο έτος, θα έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε και φιλόδοξους στόχους για τον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα και θα κληθούμε να συζητήσουμε την κατανομή των κονδυλίων. Στη συζήτηση λοιπόν για τη μελλοντική ΚΑΠ δεν μας υποχρεώνει κανείς να τηρήσουμε πλέον ανώτατα όρια για τον πρώτο και δεύτερο πυλώνα. Θα χρειαστούν νέες ε, ισορροπίες για τις άμεσες ενισχύσεις και για τους φιλόδοξους στόχους στο δεύτερο πυλώνα. Αλλά όλα αυτά φυσικά θα γίνουν μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαίρομαι λοιπόν που έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε μια νέα κατανομή. Και να είστε σίγουροι ότι στα πλαίσια του σώματος του, των Επιτρόπων θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα επιχειρήματα για να καταλάβουν και οι συνάδελφοι γιατί είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια αποτελεσματική αγροτική πολιτική. Προκειμένου να έχει και το σωστό προπολογισμό η πολιτική αυτή και παρουσιάσαμε τα σχετικά επιχειρήματα που υποστηρίζουν αυτή τη θέση και βλέπουμε πως έχει η κατάσταση στην αγορά δεδομένης και της ρευστότητας των τιμών, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα στην παγκόσμια αγορά. Να είστε βέβαιοι λοιπόν ότι συνειδητοποιώ ότι υπάρχει αυτή η ευθύνη τώρα για τις ορεινές περιοχές και για τις μειονεκτικές περιοχές. Θα πρέπει να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με το θέμα αυτό, όχι μόνο για να διατηρηθεί απαραίτητα η γεωργία στις περιοχές αυτές, αλλά προκειμένου η ειδική αυτή παραγωγή να χρησιμοποιηθεί, να αξιοποιηθεί. Και προς αυτήν την κατεύθυνση φυσικά θα ασχοληθώ ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Δεύτερη ερώτηση. Νομίζω ότι δείξατε ότι ξέρετε ποιες είναι οι μελλοντικέ προκλήσεις στην αγροτική πολιτική. Σας συγχαίρω γι' αυτό, αλλά να μην ξεχνάμε ότι το θεμέλιο της γεωργικής πολιτικής είναι ο ίδιος ο γεωργός και αντιμετωπίζουμε τη γύρανση του πληθυσμού. Ποια μέτρα θα προτείνετε για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα αυτό και ποιες προοπτικές θα ανοίξετε για τους νέους ε, αγρότες, ο Επιτροπός. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους είπα ότι η πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου θα πρέπει να παραμείνει στα πλαίσια της αγροτικής πολιτικής, γιατί εκεί μπορούμε να βρούμε λύσεις για όσους ε, ζουν και θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται στην Ήπεθρο και για τους αγρότες. Και νομίζω ότι όλα αυτά είναι αλληλοσυνδεόμενα. Μπορούμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη της Ήπεθρου μαζί με την ανάπτυξη την γεωργική. Αν είναι ανεπτυγμένη σωστά η Ήπεθρος, αυτό σημαίνει ότι είναι σωστή και η ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης και νομίζω ότι ναι, νέοι αγρότες είναι πολύ σημαντικός ε, παράγοντας γιατί το δημογραφικό πρόβλημα είναι σημαντικό. Και σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις έχω ιδιαίτερα υπόψη μου τους νέους γιατί και αυτοί χρειάζονται επενδύσεις για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των εκμεταλλεύσεων και το γνωρίζω αυτό, είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει και στην Ρουμανία. Είναι απαραίτητη η σταθερότητα, είναι απαραίτητη η προβλεψιμότητα και έχουμε τέτοιες δυνατότητες στον πρώτο πυλώνα. Έχουμε αυτές τις δυνατότητες και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις άμεσες αυτές πληρωμές για να ενισχύσουμε τη σταθερότητα. Ο Γκαρσία Περές. Presidente, señor candidato a comisario, he escuchado con, con agrado eh, como en reiteradas. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα με χαρά σχετικά με μια μεγάλη πρικοδότηση της ΚΑΠ. Σύμφωνο, είμαι ικανοποιημένη. Αλλά όμως είναι απαραίτητα και άλλα μέσα για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της ε, ΚΑΠ. Λοιπόν, εμείς έχουμε μεταπητική βιομηχανία και μεγάλα συστήματα διανομής που ελέγχουν τα πάντα. Και όταν οι γεωργοί προσπαθούν να διαπραγματευτούν τις τιμές τους δίνεται το επιχείρημα του ανταγωνισμού κλπ. λοιπά Εσείς θα δώσετε δυνατότητες ανταγωνιστικές στους γεωργούς μας ούτως ώστε να προβάλλουν και αυτοί τα δικά τους επιχειρήματα και να πάρουν και αυτοί τη μοίρα τους στα χέρια τους. Λοιπόν, εγώ να σας πω ό,τι θέλετε για το δικό μου χαρτοφυλάκιο. Εσείς όμως γνωρίζετε πολύ καλά ποιος είναι ο αρμόδιος επίτροπος για τα θέματα ανταγωνισμού και ποιες είναι οι αρμοδιότητές του. Αυτός λοιπόν είναι που πρέπει να βρει ειδικά μέτρα ε, για τον ανταγωνισμό στην ε, αγορά των γεωργικών προϊόντων, όχι για να εμποδίσει στην ανάπτυξη της αγοράς, αλλά για να βοηθήσει Και αυτό φυσικά μπορεί να γίνει ενθαρρύνοντας στους διεπαγγελματικούς οργανισμούς, τον διάλογο μέσα στο ίδιο το δίκτυο και εάν καταλήξουμε ότι μπορούμε να έχουμε παρεκκλήσεις ή εξαιρέσεις που θα μπορούσαν να οργανώσουν καλύτερα τη λειτουργία του δικτύου, τότε εγώ είμαι έτοιμος να συζητήσω σχετικά με τον αρμόδιο για τον ανταγωνισμό σχετικά με την προσαρμογή των κανόνων. Υπάρχουν όμως σε ευρωπαϊκό επίπεδο τεράστιες απαιτήσει ε, για τη λειτουργία της αγοράς. Για τα οποροκυπευτικά πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε μια λύση, να βουλέψει καλύτερα η αγορά. Θα ξαναπροβάλλω λοιπόν αυτά τα επιχειρήματα. Η κυρία Γκαρσία Πέρες δεν, έχει, δεν θέλει να κάνει επερώτηση. Ο κύριος Μάτο. Εσείς είπατε κύριε Επίτροπε ότι πρέπει να εγγυηθούμε το εισόδημα των γεωργών. Εγώ συμφωνώ και προσυπογράφω. Αλλά στις υπερπεριφερειακές περιοχές φυσάει κακός αέρας για τη γεωργία. Τα πράγματα πάνε πολύ άσχημα, απειλείται άμεσα η γεωργία σε αυτές τις περιοχές. Πεστε μας τι σκοπεύετε να κάνετε εσείς για να διατηρήσετε την αηφορία των υπερπεριφερειακών περιοχών της Ένωσης που έχουν ένα πρόβλημα, την μπανάνα. Η συμφωνία που κατέληξαν η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής κατέβασαν από 259 σε 199 τη τιμή της μπανάνας και αυτό θα οδηγήσει σε τεράστιες απώλειες. Τι θα κάνετε εσείς Μπορείτε να αντισταθμίσετε αυτήν την απώλεια. Στους γεωργούς δίνοντας ένα φακελάκι ας πούμε. Για τις υπερπεριφερειακές περιοχές ξέρετε ότι υπάρχει ένα ειδικό πρόγραμμα το ΠΟΣΕΗ e e, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει σε αυτές τις ε, περιφέρειες. Εμείς Μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό το πρόγραμμα και να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε και τις, ε, τις λύσεις ε, γιατί θέλω να παραμείνει η γεωργία σε αυτές τις περιοχές τώρα για τις μπανάνες πολύ καλό πράγμα αυτή η διαπραγμάτευση αυτή η συμφωνία συγγνώμη εδώ και χρόνια γινόταν διαπραγματεύσεις και υπήρχαν προβλήματα και στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων μας στην ΠΟΕ είναι πάρα πολύ καλό πράγμα. Ξέρετε όμως ότι υπάρχουν αποζημιώσεις, υπάρχει ένα σύστημα αποζημιώσεων για τους μπανανοπαραγωγούς το οποίο ήδη το έχουμε προβλέψει και θα δούμε εμείς τι περιθώρια έχουμε για να κάνουμε διορθώσεις αν φυσικά χρειάζεται και είναι αιτιολογημένο. Μα μπορεί να είναι καλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η συμφωνία, αλλά για τους κοινοτικούς παραγωγούς δεν είναι καθόλου καλή αυτή η συμφωνία, αν δεν συνοδεύεται από άλλα μέτρα. Εγώ θέλω να εγγυηθούμε το μέλλον αυτού του κλάδου. Είναι θεμελιώδης ε, ε, από περι περιβαλλοντικής ε, πλευράς η επιβίωση αυτού του ε, κλάδου και οικονομικά διότι στα Κανάρια νησιά είναι χιλιάδες οικογένειες που ζουν από την μπανάνα. Πρέπει λοιπόν να εγγυηθούμε το εισόδημα των γεωργών. Εσείς το έχετε στα χέρια σας, υπερασπιστείτε το. Σίγουρα θα, θα, θα καταλαγιάζουν κάπως τα πράγματα και θα υπάρχει μια σχετική ειρήνη με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής στον τομέα αυτό, αλλά μην νομίζετε ότι θα ηρεμήσουν οι δικοί μας Γεωργοί. Σε κοινοτικό επίπεδο ήδη έχουν δοθεί πολλά λεφτά, 250 εκατομμύρια το χρόνο για το πρόγραμμα ΠΟΖΗ. Ξέρω εγώ τι προβλήματα μπορούν να προκύψουν και βάσει της έκθεσης που θα μας κατατεθεί θα δούμε ποιο θα είναι το μέλλον αυτού του προγράμματος. Εγώ δεν μπορώ τώρα να σας δώσω νούμερα, σίγουρα θα φανταστούμε κάποια διόρθωση. Εγώ Έχω συνέστηση του προβλήματος. Ήδη έχουν δοθεί πολύ σημαντικά ποσά σε αυτές τις χώρες. Πρέπει να δούμε όμως τι περιθώριο θα έχουμε στο μέλλον. Ωραία. Ο Ούλερη. Ε, κύριε Ρόντος, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Τσιόλος. Απαντήσατε ήδη πολλά ερωτήματα και είναι δύσκολο κανείς μετά από τόσες ερωτήσεις να βρει ένα νέο θέμα, αλλά βρήκα ένα νέο θέμα. Παραγωγή δημοσίων αγαθών. Αναφέρεται πάντα ως ένας λόγος για την περαιτέρω διατήρηση της ΚΑΠ. Πέρα από την παραγωγή τροφίμων, η γεωργία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για το κοινωνικό, για την κοινωνική ευημερία, όπως για παράδειγμα την φροντίδα των πολιτισμικών τοπίων, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη διατήρηση της ποιότητας των υδάτων και του εδάφους. Τα αγαθά αυτά θα πρέπει να αποζημιώνονται με το σωστό τρόπο, προκειμένου να δημιουργούνται κίνητρα για τους αγρότες να διατηρούν αυτά τα κοινά αγαθά. Πώς θα φροντίσετε λοιπόν οι γεωργοί να συνεχίσουν να είναι πρόθυμοι να διαδραματίζουν το ρόλο αυτό και πώς φαντάζεστε ότι θα διαμορφωθεί η αποζημίωση σε ό,τι αφορά την παραγωγή αυτών των δημόσιων αγαθών. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας, κυρία Ρόντουστ. Είναι δύσκολο να βρει κανεί νέε ερωτήσει, αλλά είναι και δύσκολο για μένα να βρω καινούργιε απαντήσει. Αλλά χαίρομαι που ανταποκριθήκατε στην πρόκληση αυτή, γιατί όντω Δεν έχουμε συζητήσει ακόμα πολύ για τα δημόσια αυτά αγαθά, παρά το γεγονός ότι έχω ήδη αναφέρει ότι σημαντικό μέρος της ε, αγροτικής ανάπτυξης ξεπερνάει το επίπεδο της παραγωγής τροφίμων. Χαίρομαι λοιπόν που πολλά κράτη-μέλη έχουν προβλέψει μεγάλα κονδύλια για την προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα της ΚΑΠ και θεωρώ ότι όντως εκεί είναι ο τομέας στον οποίο θα πρέπει να βρούμε καινούριου μηχανισμούς ε, προώθησης για να προωθήσουμε αυτά τα περιβαλλοντικά αγαθά. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ε, κανόνες ε, για την πολλαπλή συμμόρφωση σε ό,τι αφορά τον κλάδο αυτό. Και αυτοί θα πρέπει να συνεχίσουν να υφίστανται, αλλά νομίζω ότι στον δεύτερο πυλώνα θα πρέπει να προωθηθεί και η κοινοτομία. Νέες ιδέες, νέες προτάσεις για την προστασία του τοπίου, των ζώων και ούτω καθεξής. Νομίζω λοιπόν ότι τα στοιχεία αυτά θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Και σίγουρα θα προσθέσουμε και σημαντικές πτυχές για την προστασία του κλίματος, γιατί φυσικά η γεωργία θα πρέπει να προσαρμοστεί και στις προκλήσεις της αλλαγής του κλίματος. Ξέρω ότι και εκεί υπάρχουν σημαντικές καινοτομικέ ιδέες, τις ανέφερε άλλωστε και ο Ζωζέ Θα πρέπει να προωθήσουμε λοιπόν τις καινοτομίες αυτές και να τις προωθήσουμε με τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Αλλά να είσαστε βέβαιοι ότι πρόκειται για ένα από τα βασικά θέματα που απασχολούν στο δεύτερο πυλώνα. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας θα πρέπει να σκεφτούμε στο δεύτερο πυλώνα, κατά καταλαβα αυτό, αλλά σας άκουσα με προσοχή τις τελευταίες δύο ώρες και έχουμε πάρα πολλά να επεξεργαστούμε στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα. Με το 11% του ΑΕΠ μας πώς πρόκειται να τα καταφέρουμε όλα αυτά. Σας ρωτώ λοιπόν, θα ταχθείτε υπέρ της ενίσχυσης του προπολογισμού στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα. Όπως σας είπα ήδη, χρειαζόμαστε έναν προϋπολογισμό ο οποίος θα ανταποκρίνεται και στις φιλόδοξους στόχους που θα θέσουμε. Και εννοείται ότι θα ζητήσω έναν προϋπολογισμό ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις φιλόδοξες αυτές στους φιλοδοξούς αυτούς τους στόχους. Και αυτό θα καθοριστεί από κοινού και με το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να βρούμε μία ισορροπία μεταξύ των ε, δημοσιονομικών μας ε, δυνατοτήτων και των φιλόδοξων στόχων μας. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που εντάσσονται στον δεύτερο πυλώνα, αλλά αυτό καταδεικνύει ακριβώς ότι δικαιολογείται ο υψηλός προϋπολογισμός για την γεωργική πολιτική και ελπίζω να καταφέρω να πείσω και τους άλλους συναδέλφους ότι χρειάζεται μια συνέχεια στον τομέα αυτό ξέρω ότι στο εσωτερικό του, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία. Αλλά δικός μου ρόλος είναι να παρέχω επιχειρήματα τα οποία θα δικαιολογήσουν την ισχυρή ΚΑΠ που χρειαζόμαστε και χαίρομαι που με υποστηρίζετε και μέσα από τις ερωτήσεις σας σήμερα. Η συνάδελφος Νεντελτσέβα έχει το λόγο. Μαρία Νεντελτσέβα. Έχεις το λόγο. Ξέρετε, Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα, μας συγχωρείτε μισό λεπτό. Problema di traduzione, adesso arriviamo chiediamo una Εντάξει, μπορείτε να συγκινήσετε. Να μιλήσω βουλγάρικα ή να μιλήσω γαλλικά τελικά. Μπορείτε να μιλήσετε στη γλώσσα σας. Σας ευχαριστώ Κύριε Επίτροπε, η ιδέα σας για ε, πιο ισότιμο καταμερισμό των άμεσων πληρωμών μεταξύ των κρατών μελών και της σχηματοδότησης των περιφερειών ε, πέσερε την προσοχή μου. Ε, εσείς εκθέσατε την δομή και τις ιδέες σας ως προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορείτε να μας πείτε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά σας. Έχετε τρόπο να κατανέμεται τα ταμεία με τρόπο αντικειμενικό. Θεωρείτε πως ε, σε ορισμένους τομείς ή για ορισμένα προϊόντα θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε το παλαιό σύστημα ενισχύσεων, όπως για παράδειγμα την ενίσχυση που δίνει τους παραγωγούς καπνών για τα ευαίσθητα δηλαδή προϊόντα. Ευχαριστώ. ο Επίτροπος. Για το χρονοδιάγραμμα. Καταρχήν έχω την πρόθεση να διοργανώσω μια δημόσια διαβούλευση και γι' αυτό ακριβώς το λόγο σας έλεγα ότι δεν επιθυμώ να ε, ε, εκφράσω και τώρα κάποιες ιδέες, θέλω πρώτα να ακούσω ε, μέσω από μια δημόσια διαβούλευση. Και βέβαια η συζήτηση με τα κράτη μέλη και με το Κοινοβούλιο θα είναι πολύ σημαντική. Κατά τη διάρκεια του 2010 λοιπόν θα ξεκινήσει αυτή η διαβούλευση με στόχο, αν είναι δυνατόν, στο πλαίσιο της ε, Κομισιόν να ολοκληρώσουμε για μια ανακοίνωση πριν το τέλος του χρόνου, πριν να προτείνουμε νομοθετικό κείμενο, μια ανακοίνωση της Επιτροπής που θα εκθέτει εν γέννη τις γιατί για την ΚΑΠ μετά από το 2013 και έπειτα το 2011 να προτείνουμε και νομοθετικό κείμενο βέβαια. Το χρονοδιάγραμμα αυτό θα εξαρτηθεί επίσης και από το χρονοδιάγραμμα των δημοσιονομικών προοπτικών διότι είναι σημαντικό όπως, σας έχω, ε, όπως έχω πει και παλιότερα να συνδέσουμε τις ε, φιλοδοξίες μας με τις ε, οικονομικές δυνατότητες, τις, τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες και Ξέρω ότι σας ανησυχούν όλα αυτά ως βουλευτές. Ε, από ό,τι σου γνωρίζω θα υπάρξει μια έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την εικόνα, για το όραμα για την ΚΑΠΑ. Ξέρω ότι ο κύριος Λάιον είναι εισηγητής για αυτό το θέμα, αν δεν κάνω λάθος. Για την αντικειμενική κατανομή και τα ευαίσθητα σημεία για τον καπνό υπάρχει μια μεταρρύθμιση που έχει αποφασιστεί από το 2004. Υπήρξε μια μεταβατική περίοδος και υπήρξε και υπάρχει ακόμα για τα κράτη-μέλη δυνατότητα για προσαρμογή μιας ειδική ενίσχυσης για τον τομέα αυτό. Αν όμως μιλάμε αυστήρα για τον καπνό και συγκεκριμένα για τον καπνό, θα πρέπει να είμαστε συνεπείς όσον αφορά τις προσδοκίες των Ευρωπαίων φορολογούμενων για το συγκεκριμένο προϊόν και φαντάζομαι πως καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλώ, αλλά επιμένω ότι τα κράτη-μέλη έχουν ακόμα περιθώριο λιγμό, έχουν τη δυνατότητα να δώσουν ειδικέ ενισχύσεις για τον τομέα αυτό. Επερώτηση υπάρχει. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ακόμη ερώτηση στην εισήγησή σας. Μιλήσατε και επιμείνατε για την διαφοροποίηση ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειες και η ΚΑΠΑ στο μέλλον θα πρέπει να επιτρέπει μια τέτοια διαφοροποίηση. Ωστόσο σήμερα ορισμένα σε ορισμένα κράτη-μέλη το κόστη παραγωγής είναι εξαιρετικά υψηλά, πράγμα που οφείλεται στις ε, κλιματικές συνθήκες. Για να υπάρχει τώρα καλύτερη παραγωγή, πώς μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας την, την βόρεια, την σκανδιναβική ιδιαιτερότητα, ας πούμε, για τον προπολογισμό 2013 και μετά το 2013 και πώς ε, βλέπετε πώς θα μπορέσουμε μάλλον να βρούμε λύσεις στα πολύ ιδιαίτερα προβλήματα κάποιων περιφερειών της Ευρώπης και ταυτόχρονα να αγγιηθούμε τα συμφέροντα όλων. Εφόσον τα συμφέροντα όλων των γεωργών. Υπάρχουν βεβαίω διαφορέ ανάμεσα στι ε, περιφέρειες και αυτέ οι διαφορέ λαμβάνονται υπόψη σήμερα ήδη μέσω των ειδικών μέτρων της πολιτικής ανάπτυξης της υπαίθρου που ε, στόχο έχουν ε, ακριβώς αυτές τις περιοχές. Έχω ότι θα πρέπει να έχουμε μια τάση ισότητας και δικαιοσύνης στο πλαίσιο των άμεσων πληρωμών και αναφερόμουν σε αυτές τις τάσεις γιατί για ορισμένε περιοχές θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κάποιες ιδιαιτερότητες προσέγγισης αλλά και ε, υπολογισμού ώστε να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε τον ιδιαίτερο τους χαρακτήρα. Εκεί δηλαδή όπου η παραγωγικότητα επηρεάζεται από τις κλιματικές ε, συνθήκες, ε, ισορροπημένη κατανομή της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια μέσω της αντίληψης των κριτηρίων της κατανομής των αμέσων πληρωμών αλλά και μέσω ειδικών εργαλείων που έχουμε στο πλαίσιο της ε, πολιτικής ε, ανάπτυξης υπαίθρου από την άλλη πλευρά νομίζω πως θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις για να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιφέρειας. Ωραία, τώρα το λόγο έχει η κυρία Αντάντσιλα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τσόλος. Ποια είναι τα ιδιαίτερα μέτρα τα οποία προβλέπετε για να μειωθεί η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα νέα και τα παλιά κρατημέλη, ώστε να αυληθούν τα προβλήματα των τελευταίων, ώστε να αναπτύξουν μια ανταγωνιστική γεωργία που θα μπορεί να σταθεί και σε διεθνές επίπεδο και για να πάψει η μετακίνηση των γεωργικών πληθυσμών προς τις πόλεις που δημιουργεί ε, δημογραφικές, ε, δημογραφικά προβλήματα. Κυρία Τανσίλα, όπως έχω ήδη υπογραμμίσει, για το μετά το 2013 έχουμε στη διάθεσή μας ε, στοιχεία και κριτήρια που μας επιτρέπουν να ξεκινήσουμε από μια νέα βάση για την κατανομή των ενισχύσεων και από αυτή την άποψη μπορούμε να λάβουμε υπόψη τα στοιχεία τα οποία αναφέρατε στα νέα στοιχεία, στα νέα κράτη-μέλη, συγγνώμη, ε, όπως και στη Ρουμανία, βρισκόμαστε στη φάση της ανάπτυξης, της μεγέθυνσης ε, του επίπεδου των ενισχύσεων και νομίζω πως αυτό το χρόνο ή στο διάρκεια του επόμενου χρόνου θα τελειώσει το πρόγραμμα αυτό λόγω των νέων κριτηρίων κατανομής των ενισχύσεων. Τέλος, ε, μάλλον στη συνέχεια για να δοθεί τέλος στην αγροτική έξοδο. Έχουμε πολύ σημαντικά προγράμματα και εδώ νομίζω πως μπορούμε να βρούμε και ειδικέ προβλέψεις. Υπάρχουν οι άμεσες πληρωμές οι οποίες θα κατανεμηθούν με βάση πιο ισότιμα κριτήρια από ό,τι μέχρι σήμερα. Ε, ε, αυτό θα γίνει και με βάση τα ε, την εθνική μας κλίμακα όπου θα πρέπει να βρούμε μια, ένα μείγμα ανάμεσα στις άμεσες πληρωμές αλλά και τις δυνατότητες που προφέρονται από τον εξυγχρονισμό της γεωργίας. Η κυρία Τανσίλα δεν θέλει να υποβάλει επερώτηση. Ωραία, περνάμε άμεσα στο κύριο Κλάτφερτ. Φέλτερ. Σας ευχαριστώ σε τελική ανάλυση είναι δύσκολο στο τέλος να βρει κανείς όντως ε, καινούργιες ερωτήσεις, γιατί έχουν τεθεί πάρα πολλά σχετικά ερωτήματα, αλλά ε, αξιολογήσαμε κάποιες από τις απαντήσεις σας ε, και μου άρεσε αυτό που αναφέρατε για την διατήρηση των αξιών της ΚΑΠ και ότι θα απορρίψετε την επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ. Και χαίρομαι που θα καταβάλλετε προσπάθειες για να προστατεύσετε τους Ευρωπαίους αγρότες από τις τρίτες χώρες. Και σε ό,τι αφορά τις πολύ αυστηρούς όρους για την προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι είδους μέτρα θα λάβετε για να γίνουν επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης, προκειμένου να μειωθούν στη γεωργία και η εκπομπή του εξουδίου του άνθρακα. Για τις ενεργειακές εξοικονομήσεις μιλήσατε. Το θέμα είναι αυτό λοιπόν. Ο εξυγχρονισμός των αγροτικών τεχνολογιών θα λάβει υπόψη τη διάσταση αυτή. Αυτό θα γίνει είτε μέσω των εθνικών σχεδίων για την ανάπτυξη της υπέτρου, είτε των μέσων στο δεύτερο πυλώνα. Άρα αφενός έχουμε τη δυνατότητα να προωθήσουμε νέες τεχνολογίες και σε ό,τι αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας. Και ξέρω ότι υπάρχουν και επενδυτικά προγράμματα τα οποία αποσκοπούν στην ε, ανάπτυξη τέτοιων νέων τεχνολογιών και όπως σας είπα ότι με τη, συνεργασία της Γενικής Διεύθυνσης ε, έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η ενεργειακή, η αξιοποίηση των τεχνολογιών αυτών στην αγορά. για την προώθηση και δημοσίων αγαθών. Και φυσικά σε αυτά τα δημόσια αγαθά συγκαταλέγεται και η μείωση του διοξυδίου του άνθρακα. Άρα θα υποστηρίξουμε τέτοιες καινούργιες ιδέες καινούργιες προτάσεις. Ίσως να μην υπάρχει κοινωτικός ε, μηχανισμός προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί υπάρχουν πολλές και διαφορετικές καταστάσεις και τάσεις σε τοπικό επίπεδο. Και θα πρέπει εμείς να διασφαλίσουμε ότι η γεωργία σε εθνικό και τοπικό επίπεδο θα χρησιμοποιεί αυτές τις τεχνολογίες και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα των μέσων αυτών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ. Στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, στη χώρα μου, δεν υπάρχει δυνατότητα να δαπανηθεί ούτε ένα ευρώ από το δεύτερο πυλώνα για την μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί προσοχή στο θέμα αυτό, προκειμένου και τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν τέτοια προγράμματα. Και θα πρέπει να φροντίσουμε τις νέες ε, ρυθμίσεις, τις νέους ε, κανονισμούς, γιατί κάποιοι κανονισμοί θα προκαλέσουν δυσκολίες στους ε, γεωργούς. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, των ζέων. Όλα αυτά ενδεχομένως να μειώσουν την αποδοτικότητα και να αυξήσουν και την ενεργειακή κατανάλωση αλλά και τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Πώς θα αντιμετωπίσετε τέτοιο ενδεχόμενο. Απάντηση. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα μέσα του δεύτερου πυλώνα, τα κράτη-μέλη έχουν περιθώριο ελιγμού σε ό,τι αφορά την θέση των προτεραιοτήτων του σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Για το διάστημα μετά το 2013 θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι και ο σχετικός κανονισμός θα περιλαμβάνει πιο συγκεκριμένες διατάξεις. Αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο της κοινή αγροτικής πολιτικής. Και ο σκοπός αυτός για τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα είναι πολύ σημαντικός και για όλη την ευρωπαϊκή πολιτική. Τώρα, για τις ε, απλές ρυθμίσεις και για την έλλειψη αντιφάσεων μεταξύ της προστασίας των ζώων και της προστασίας του περιβάλλοντος και το καθεξής. Εδώ πέρα χρειάζεται προσοχή. Στο σημείο αυτό, στη συζήτηση, φυσικά θα πρέπει να προκύψει και μια ισορροπία ως προς την ενεργειακή κατανάλωση, αλλά σε ό,τι αφορά τα θέματα προστασίας των ζώων, πρόκειται για διατάξεις οι οποίες θα πρέπει να διατηρηθούν, γιατί αποτελεί φυσικά σημαντικό θέμα αυτό. Μάλιστα και τώρα περνάμε στον Τζοβάνι Λαβία. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, να σας ευχαριστήσω καταρχήν για όλα όσα μας είπατε σήμερα το πρωί, διότι δώσατε ορισμένα στοιχεία ε, πολύ ενδιαφέροντα και αξιόλογα για τα μέλη αυτής της Επιτροπής. Και σε άλλες όμως ακροάσεις και σε αυτές δηλαδή του τρόπου για τον προϋπολογισμό δεν ακούστηκε τίποτα για την μείωση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ. Κανένας λοιπόν δεν έδωσε κάτι το βάσιμο για την ύπαρξη αυτή του μη εγγράφου. Και ρωτώ εγώ λοιπόν, εμείς υποστηρίζουμε την γεωργική πολιτική και τους διάφορους κλάδους της. 16% αυτό ας πούμε παίρνουν τα οποροκυπευτικά και είναι το 4% των ενισχύσεων. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν πώς θα αντιμετωπίσετε εσείς την χρηματοδότηση της Μεσογειακής Γεωργίας και πώς θα την ενισχύσετε αναλογικά με τα υπόλοιπα προϊόντα. Βεβαίως, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη βαρύτητα του κάθε τομέα και αν κάνουμε μία σύγκριση των επιδοτήσεων σίγουρα θα μπορούμε να διαπιστώσουμε ανισορροπίες για τα όποροκυπευτικά η προσοχή μας θα πρέπει να δοθεί στη διαμόρφωση ενός μηχανισμού που θα διασφαλίζει την ισορροπίες. Η μεταρρύθμιση της αγοράς των οποροκυπευτικών μας προσφέρει τα απαραίτητα μέσα η χρηματοδότηση σε εθνικά πακέτα στα κράτη-μέλη επιτρέπει ε, στα κράτη να βρίσκουν τις ε, λύσεις ε, για τη χρηματοδότηση των διαφόρων προϊόντων. Εγώ ως επίτροπος θα πρέπει να βρω μια ισορροπία μεταξύ των διαφόρων τομέων και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όχι μόνο τη βαρύτητα του τομέα αλλά και την ιδιαιτερότητά του. Για τα οποροκυπευτικά έχουμε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία δεν μπορούν να ισχύσουν για άλλα προϊόντα. Εγώ δεν μπορώ να σας υποσχεθώ τίποτα λέγοντας ορίστε ε, το χ ο για τον ύψιλον τομέα. Όχι για τον κάθε τομέα πρέπει να βρούμε την ιδιαιτερότητά του. Κατά την ακρόαση ακούσαμε πολλές φορές να αναφέρεστε για την παρέμβαση στην αγορά ε, σε μοντέλα αντίστοιχα με αυτά των όπορο πέρα από την ενίσχυση του 4,1 της αξίας της παραγωγής υπάρχει και ένα 0, κάτι της εκατό για τις παρεμβάσεις στην αγορά. Όμως τα τελευταία χρόνια αυτός ο μηχανισμός για τα οποροκυπευτικά πρέπει να διορθωθεί, να τακτοποιηθεί. Εγώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σημειώνω και το βλέπω και με καλό μάτι αυτό που λέτε να επεκταθεί η μέθοδος των οποροκυπευτικών και σε άλλα προϊόντα. Αλλά όμως τονίζω ότι υπάρχει και η ανάγκη να προσαρμοστεί αυτός ο μηχανισμός στις ισορροπίες της αγοράς που όλοι θέλουμε. Αυτός ο ειδικό μηχανισμός για τα ποροκυπευτικά είναι πρόσφατος. Εδώ και ένα χρόνο έχει αρχίσει, αν δεν κάνω λάθος, να ισχύει. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πολύ νωρίς να ανασύρουμε συμπεράσματα για το κατά πόσο αυτός ο μηχανισμός είναι αποτελεσματικός και κατά πόσο θα πρέπει να διορθωθεί ή όχι. Ξέρω όμως ότι στα διάφορα στάδια προβλέπεται μία ανάλυση αποτελεσματικότητας του συστήματος και όταν θα έχω επαρκή στοιχεία και εμπειρία για αυτόν τον μηχανισμό είμαι έτοιμος να τον επανεξετάσω. Θεωρώ όπως, ε, όμως ότι ε, έχουμε μία καλή αφετηρία στον τομέα αυτό. Κυρία Μαγκίνε. Ευχαριστώ πρόεδρε κύριε υποψήφια Επιτροπετρία. Σχόλια να σας ε, συγχαρώ για την έμφαση που δίνετε στην ασφάλεια των τροφίμων και να σας καλέσω στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζω να επικυρωθεί προκειμένου η Επιτροπή να επικεντρωθεί στην ασφάλεια των τροφίμων όχι μόνο όταν αυξάνονται οι τιμές αλλά και όταν πέφτουν οι τιμές για τους παραγωγούς. Και κατά δεύτερον να σας καλέσω να έρθετε σε επαφή με την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και να τονίσετε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ σούπερ μάρκετ και παραγωγών και επίσης να μιλήσετε σε θέματα επιστημονικά όπου Παριγράφατε η σχέση της κοινωνίας με τους γενικατικά τροποποιημένους οργανισμούς για τους τροπολογισμούς. Θα είναι δύσκολες οι συζητήσεις. Θα μπορούσατε να σχολιάσετε και να μου πείτε ειλικρινά για να τη μεταβιβάσουμε στους γεωργούς μας η ανακατανομή που θα γίνει μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ των περιφερειών των κρατών μελών και μεταξύ των γεωργών. Πώς ε, θα μεταχειριστούμε σε αυτή την εξίσωση τους χαμένους και τους κερδισμένους και θεωρείτε ότι θα μετατοπιστεί η περίοδος αναφοράς, θα μετατοπιστεί προς, το, προς τα μπροστά ή θα μείνει στο παρόν ιστορικό πλαίσιο. Απάντηση. Θα σας απαντήσω ανοιχτά. Όσο πιο ανοιχτά μπορώ στην παρούσα φάση. Είπα ήδη ότι το ιστορικό πεδίο αναφοράς, πλαίσιο αναφοράς, δεν αποτελεί πλέον μία βιώσιμη λύση για το μέλλον. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την πολυμορφία που υπάρχει και υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Δεν μπορούμε να επανέλθουμε σε κάποιους μηχανισμούς ρύθμισης της αγοράς που είχαν θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία της αγοράς και όπως σας είπα αυτό το ιστορικό πλαίσιο πλέον ανήκει στην ιστορία, στο παρελθόν. Χρειαζόμαστε νέες λύσεις. Τώρα, το ποια θα είναι τα ποσά τα οποία θα πρέπει να ανακατανεμηθούν μεταξύ των κρατών μελών και των ε, περιφερειών. Δεν μπορώ να σας πω οτιδήποτε σήμερα. Όχι επειδή δεν θέλω, αλλά επειδή πρώτα πρέπει να γίνει συζήτηση. Αυτό που θα γίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να ε, καταρτιστούν όσο το δυνατόν πιο ισορροπημένα κριτήρια και σήμερα είδαμε πόσα συγκεκριμένα προβλήματα ανακύπτουν σε διάφορες περιοχές, περιφέρειες και στα διάφορα Αυτό που είναι σημαντικό είναι το εξή ωστόσο. Βρισκόμαστε στη φάση της συναπόφασης και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο διάλογος. Θα συζητήσουμε λοιπόν τέτοια θέματα και γι' αυτό εκτιμώ την αρμοδιότητα της Επιτροπής σας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χρειαζόμαστε ισορροπημένες λύσεις για μια Ευρώπη της πολυμορφίας. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο Μαγκίνες, ε, επερώτηση. Μια περίεργη ερώτηση. Δεν ξέρω τι σε προτιμάτε στη μουσική. Σας αρέσουν οι Beatles ή ο Paul McCartney ειδικότερα. Αλλά θα προασπιστείτε τους παραγωγούς, ε, τους εκτροφείς ε, ζώων στην Ευρώπη από επιθέσεις όπως αυτές του Πολ Μακάρτνη και θα εγγυηθείτε στο Κοινοβούλιο ότι θα προασπίσετε αυτές τις ιδέες σε ευρωπαϊκό ιδέα, στο ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί σε πολλές περιπτώσεις κάποιες τρελές και χαζές ιδέες ε, πιάνουν ρίζες αν δεν τις ε, καταπολεμήσουμε αμέσως. Απάντηση. Ναι, εννοείται. Ασφαλώς μου αρέσει και η μουσική του Πολ Ο καθένας μπορεί να έχει τις δικές του απόψεις και αξίες για τα θέματα αυτά και σέβομαι τις απόψεις κάθε ατόμου, αλλά για αυτό που είπατε. η πιο αποτελεσματική και σωστή πολιτική στάση μπορεί να διαμορφωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ ως Επίτροπος για τη Γεωργία μπορώ να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να υποβάλω ισορροπημένες προτάσεις, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη διάφορες ε, πραγματικότητες, διάφορα χαρακτηριστικά, προτάσεις ε, για την αξιοποίηση των προϊόντων των αγροτών. Τώρα, το τι θα κάνει το κάθε άτομο εξαρτάται από το ίδιο το άτομο και δεν πρόκειται να τοποθετηθώ από αυτού περαιτέρω. Ευχαριστώ. Ε, il turno... Τελειώσαμε το γύρο των ε, ονομαστικών ερωτήσεων και θα δώσω τώρα το λόγο σε ορισμένους βούλευτες διότι η σοσιαλιστική και δημοκρατική ομάδα εξοικονόμησε μερικά λεπτά στις τοποθετήσεις της όπως επίσης και η Άλντε. Ο κύριος Λεμίτσιτζακ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της ανάπτυξης της υπέτρου. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ως πρώην Υπουργή Γεωργίας σε νεα κρατημέλη, ότι τα πιο πολλά χρήματα δαπανούνται στην ε, βελτίωση της αποδοτικότητας πολλών εκμεταλλεύσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να διτηρηθεί μια ισορροπία. Δεν θα πρέπει να το διορθώσουμε αυτό, δηλαδή. Δεν θα πρέπει να παραχθεί αυτό άμεσα στους ε, αγρότες για την ενίσχυση της παραγωγής, προκειμένου να ενισχύσουμε μια δραστηριότητα η οποία έχει σταματήσει πλέον την ανάπτυξη της υπαίθρου για να ενισχύσουμε τον κόσμο που ζει στην Ήπεθρο, παρέχοντας καλύτερη ποιότητα κοινοφελών υπηρεσιών προς αυτούς. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, θεωρώ, σήμερα, η πρόσβαση στην ε, σύγχρονη υποδομή, στις σύγχρονες υποδομές. Είτε πρόκειται για εκπαίδευση, είτε πρόκειται για αθλητισμό, είτε πρόκειται για θέματα υγείας, πολιτισμού και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να αποτελέσει μια προτεραιότητα στο πρόγραμμα για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι εντελώς ξεχωριστό ως προς την διαχείριση του σκέλους αυτού. Απάντηση. Ναι, καταλαβαίνω ποια είναι η θέση σας. Ξέρω ότι είσαστε από ένα κράτος μέλος ε, της Ανατολικής Ευρώπης όπου υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα. Με την ιδιότητά μου ως Επίτροπος θα πρέπει να λάβω υπόψη πολλά και διαφορετικά προβλήματα. Υπάρχουν περιφέρειες όπου ο αριθμός των αγροτών είναι πιο περιορισμένος από ό,τι στην Πολωνία και εκεί είναι σημαντικό πέρα από την γεωργία να αναπτυχθούν και άλλες δραστηριότητε στον τομέα της υπαίθρου. Και γι' αυτό υπάρχει άλλωστε και αυτό το περιθώριο αλληγμού των κρατών μελών μέσα από τα προγράμματα ανάπτυξη τη υπέτρου, τα οποία θα καταρτιστούν σε εθνικό επίπεδο και σε κάποια κρατημέλη και σε περιφερειακό μάλιστα επίπεδο, για να ληφθούν υπόψη αυτές οι ιδιαίτερες καταστάσεις. Αυτό που περιγράψατε είναι η καλύτερη κατανομή των μέσων για διάφορες επενδύσεις, για διάφορους τομείς. Η Πολωνία ως κρατός έχει τη δυνατότητα αυτή κατά την κατάρτιση του εθνικού προγράμματός της να ορίσει συγκεκριμένες προτεραιότητες. Αλλά από, πλευρά, από πλευράς προοπτικής είναι, σημαντικό είναι να δημιουργήσουμε μηχανισμούς προκειμένου να υπάρχει αυτή η δυνατότητα κατάρτισης ε, ξεχωριστών εθνικών προγραμμάτων. Και αν θεωρείτε ότι υπάρχουν και άλλες ιδέες οι οποίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν για την πολιτική, για τον τομέα της ανάπτυξης της υπαίθρου και σε ό,τι αφορά την μεταρρύθμιση της, ε, του κανονισμού, Είμαι ανοιχτό σε προτάσεις προκειμένου να δοθεί, όπως είπα, και να εγγυηθούμε αυτό το περιθώριο ελιγμού στα κράτη-μέλη για την διαμόρφωση των προγραμμάτων τους. Μάλιστα, ο κύριος... Ο... Κυρία Πάλτσον, για ένα λεπτό. Den blivande kommissionärens föreställning om att vi kommer att få θα ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο σε σχέση με το Κύριε Πρόεδρε, και κύριοι συνάδελφοι, κύριε υποψήφιο Επιτροπέ, καταλαβαίνω πολύ καλά ότι προσπαθούμε να διατηρήσουμε αυτή τη συζήτηση και να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με κάποιους προποθέσει. προϋποθέσεις. Να διατηρήσουμε δηλαδή τον προπολογισμό που έχουμε αυτή τη στιγμή, όμως το υπόλοιπο της Ευρώπης ε, διανύει μια πολύ, ε, πολύ προχωρημένη και βαθιά κρίση. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν Πώ θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί η ΚΑΠ με μια κατάσταση προπολογισμού πραγματικά μειωμένου. Nu știu, o să vedem care este ideea, abordarea colegiului Comisiei în discuțiile care vor veni. Încă comisia, această comisie încă... Κοιτάξτε, Η Επιτροπή μας δεν έχει ακόμα αργήσει τη θητεία της, δεν έχει αναλάβει ακόμα τα καθήκοντά σου. Της, εγώ σας εξέφρασα τις απόψεις μου για τον προπολογισμό. Έχω τη συνείδηση ότι ως μέλος της Επιτροπής Μπαρόζο 2 ε, γνωρίζω πολύ καλά πως η Γεωργία χρειάζεται χρηματοδότηση. Έχουμε φιλοδοξίες που στηρίζονται από τα κράτη-μέλη και πρέπει αυτά να στηριχθούν σε δημοσιονομικό επίπεδο. Αλλά εγώ ως Επίτροπος της Γεωργίας θεωρώ πως είναι ρόλος μου και καθήκον Λοιπόν μου να ε, ε, βρω τα, επιχειρήματα που ε, οδηγούν στην, που αποδεικνύουν μάλλον την ανάγκη μια συνεπούς γεωργικής πολιτικής. Θα δώσω τώρα το λόγο. Την κυρία Ντελάγκα, ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Στα λανδικά λέμε ότι εδώ έχει κανείς δίκιο δεν σημαίνει ότι το βρίσκει και το δίκαιο του πάντα. Νομίζω ότι ξέρω και καταλαβαίνω ότι ξέρετε τι γίνεται στην πράξη για την ε, ΚΑΠ. Το θέμα όμως είναι να έχει κανείς την εξουσία να τα περάσει αυτά που ξέρει. Σας ρωτώ λοιπόν, με ποιο τρόπο θα πείσετε τους συναδέλφους σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι όλα αυτά που μας είπατε σήμερα μπορείτε να τα πραγματοποιήσετε, να τα υλοποιήσετε, δηλαδή για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική με ένα σημαντικό προπολογισμό. Πώς θα πείσετε τους συναδέλφους σας το σώμα των επιτρόπων ότι χρειάζεται αυτό. Και δεύτερη ερώτηση, πολλές φορές ε, σαν ε, ως Ευρωπαίος Επιτρόπος ε, καλείται κανείς να αναλάβει δράση κατά του κράτους μέλους από το οποίο προέρχεται και ίσως αυτό σημαίνει ότι θα υποστεί κανείς πιέσεις για να δράσει διαφορετικά. Πώς ε, θα αντιδράσετε στις πιέσεις τις οποίες αδιαφυσβήτητα θα δεχτείτε από, το, από τη χώρα σας για να ανταποκριθείτε στα καθήκοντά σας. Απάντηση πώς θα πείσω τους συναδέλφους μου πώς θα προσπαθήσω να πείσω τους συναδέλφους μου μάλλον. Ελπίζω ότι θα το καταφέρω όπως ελπίζω ότι κατάφερα να πείσω και εσάς ότι χρειαζόμαστε μια ισχυρή ΚΑΠ. Αν και φυσικά τα πράγματα εδώ ήταν λίγο πιο εύκολα από ότι θα είναι μεταξύ των συναδέλφων μου. Υπάρχουν πολύ ισχυρά, πολλά ισχυρά επιχειρήματα για την ε, ενίσχυση της ΚΑΠ. Αλλά είναι σημαντικές και άλλες πτυχές. Η πολιτική αυτή δεν μπορεί να διαμορφωθεί μία φορά και για πάντα. Θα πρέπει να δίνονται καθημερινοί αγώνες. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η παραγωγή των τροφίμων, να αντιμετωπιστούν οι κρίσεις και όλα αυτά αναζητούν, ε, ζητούν μάλλον και την δική μας παρέμβαση. Ελπίζω να σας έπεισα. Τώρα, είμαι Ευρωπαίος υποψήφιος ε, επίτροπος και αν ε, επικυρωθεί ο διορισμός μου, θα είμαι Ευρωπαίος Επίτροπος. Θα εφαρμόσω λοιπόν με αυστηρό τρόπο τους κανόνες και σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των προϋπολογισμών. Το θέμα λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα σωστά μέσα, τα οποία και μετά θα πρέπει να ελεγχθούν. Θα πρέπει να βρούμε λύσεις για να αγγίθουμε τη σωστή χρήση των μέσων, αλλά από πλευράς ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σκοπεύουμε να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη. Κομισάριο. Κομισάριο, σε λέει rinuncia suoi 5 minuti finali. Επίτροπε, αν ε, δεν θέλετε τα τελικά σας πέντε λεπτά, μπορούμε να επιτρέψουμε ακόμα κάποιες μονόλεπτες ερωτήσεις. Επιλέξτε εσείς, Επίτροπε, τι προτιμάτε. Εγώ θα μείνω πιστό σε αυτό που είπα, ότι δηλαδή ο διάλογο είναι πάρα πολύ σημαντικό και τα συμπεράσματα που θα μπορούσε κανεί να βγάλει από τα όσα είπα ε, είναι πιο σημαντικά αν συνεχίσουμε το διάλογο. Ωραία λοιπόν, μερικέ ακόμα ερωτήσει Ε, μονόλεπτες. Ο κύριο Δανέλης δεν είναι εδώ, οπότε... Α, παρακαλώ, Λουίς. Εγώ ήθελα να κάνω μία ερώτηση στο Προεδρείο. Μία έκκληση στο Προεδρείο με την έννοια ότι δηλαδή η σοσιαλιστική μας ομάδα κάναμε μία μεγάλη προσπάθεια να μην επαναλαμβάνουμε τη δεύτερη ερώτηση, την επερώτησή μας ώστε και άλλοι να μπορέσουν να πάρουν το λόγο. Και θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να αναγνωρίσετε αυτή μας την προσπάθεια και να διευρύνετε όσο γίνεται περισσότερο αυτό το διάλογο στα λεπτά που απομένω. Βεβαίως και το σέβομαι και θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντανέλης για ένα λεπτό ευχαριστώ Πρόεδρε, εδώ είμαι. Πιστεύετε ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο γεωργίας εκφράζει τις κοινέ αξίες και αρχές στις οποίες βασίζεται η ευρωπαϊκή γεωργία. Εάν ναι, ποια θεωρείτε ότι είναι τα μη διαπραγματεύσιμα του στοιχεία, εάν όχι τι μεταβολές θα προτείνατε και βεβαίως με ποιο τρόπο θεωρείτε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας μπορεί να το επηρεάσει. Ευχαριστώ πολύ. εγώ το είπα ήδη, πιστεύω ότι το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο βασίζεται καταρχήν στην ποιότητα και στη διαφορετικότητα των προϊόντων που προσφέρουμε. Όπως επίσης ε, και στη σημασία που προσδίδουμε ότι η Γεωργία θα πρέπει να παραμείνει σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυναμικά στις, σε όλες τις περιοχές και περιφερείς λαμβάνοντας υπόψη και το κοινωνικό μοντέλο της κάθε περιοχής. Διότι εμείς θέλουμε να παραμείνουν οι γεωργοί ενεργοί σε όλη την επικράτεια. Στην μελλοντική ΚΑΠ θα κοιτάξουμε να ενισχύσουμε αυτήν την άποψη. Αυτός ο δεσμός πρέπει να παραμείνει όταν μιλάμε και για διαφορετικότητα, όχι μόνο διαφορετικότητα των τροφίμων αλλά και του τύπου γεωργίας. Αυτή είναι μία από τις αξίες της ευρωπαϊκής γεωργίας και είναι ένα στοιχείο μέσα από το οποίο μπορούμε να δικαιολογήσουμε και τη χρηματοδότηση που δίνει η κοινωνία στη γεωργία. Ωραία. Ο κύριος Φάιμοντ, για ένα λεπτό. Ε, ε, θα ήθελα να καλωσορίσω το γεγονό ότι είστε επίτροπο από νέο κράτο μέλο και θα ήθελα να σα ρωτήσω για το, για το μέλλον τη γεωργική πολιτική. Η ΚΑΠ είναι κάτι πολύ διαφορετικό στα νέα κρατημέλη από ό,τι στα παλιά κρατημέλη. Είναι στόχο σα τα επόμενα πέντε χρόνια να επιτύχετε τους, τις όρου ε, σε ολόκληρη την Ένωση και θα εργαστείτε προς αυτό το στόχο, θα υποβάλλετε τις σχετικές προτάσεις, ώστε οι γεωργοί στα νέα κρατημέλη να δουλεύουν με τους ίδιους όρους όπως και οι συνάδελφοί τους στα παλιά κρατημέλη. Ευχαριστώ. Ναι, αναφέρεστε στις άμεσες πληρωμές και στον τομέα αυτό σας επιβεβαίωσα ότι θα κάνουμε προτάσεις ώστε να μην υπάρχουν πλέον διακρίσεις ανάμεσα στα παλιά και στα νέα κρατημέλη. Για τα διάφορες προσεγγίσεις ανάμεσα στον πρώτο και δεύτερο πυλώνα πιστεύω πως η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτή την ιδιαιτερότητα και άρα στο μέλλον η ΚΑΠ θα πρέπει να δώσει τα μέσα στα κράτη-μέλη ώστε να μπορέσουν με τη σειρά τους να ασχοληθούν και να αντιμετωπίσουν με ιδιαίτερο τρόπο την γεωργία. Γιατί σε πολλά κράτη-μέλη πρέπει να γίνουν περισσότερες επενδύσεις από ό,τι στα παλιά κράτη-μέλη. Και όσον αφορά τις άμεσες πληρωμές, νομίζω πως πρέπει να επιτύχουμε αυτή την ισότητα όσον αφορά τον τρόπο παροχής, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το ιστορικό κριτήριο. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Κρίσταλ Σάλντεμος. Εδώ είμαι. Να σας ρωτήσω το εξής. Η κυρία Φίσορ Μπέλ είχε υποστηρίξει μία γραμμή κατά των κρατών μελών που είχαν προβλήματα για τις άμεσες ε, επιδοτήσεις, τις άμεσες ε, πληρωμές και είχε αναστείλει μάλιστα τις άμεσες αυτές τις πληρωμές και τώρα στην ε, τελευταία έκθεση προκύπτει ότι το σύστημα αυτό λειτουργεί, αλλά κάποιες χώρες έχουν προβλήματα, μεταξύ άλλων και η Ρουμανία. Τι θα κάνετε για τη σωστή χρήση των πόρων αυτών. Απάντηση. Ναι, το ανέφερα αυτό ήδη. Αυτό που θεωρώ ότι είναι σημαντικό είναι ότι είμαστε σε θέση να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε σωστά τα μέσα και να ασκήσουμε έλεγχο για την κατανομή των πόρων. Υπάρχουν διάφορα μέσα και μέτρα με τα οποία μπορούμε να επισημάνουμε στα κράτη-μέλη ότι υπάρχουν προβλήματα. Το clearance of accounts, για παράδειγμα. Εκεί έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε ποινές όπου αυτό είναι απαραίτητο. Σε ό,τι αφορά τη Ρουμανία θα ήθελα να πω το εξής. Είμαι υποψήφιος επίτροπος πλέον και ελπίζω να εγκριθεί ο διορισμός μου. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πάρα πολύ ικανή σε ό,τι αφορά τέτοια θέματα και αυτά έχει αποδειχτεί σε ό,τι αφορά και το χαμηλό ποσοστό σφαλμάτων σε ό,τι αφορά την Ήπεθρο. Θα δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη στην αντιμετώπιση των δομικών αυτών προβλημάτων. Σας διαβεβαιώ ότι ως Ευρωπαίος Επίτροπος, θα δράσω μάλλον ως Ευρωπαίος Επίτροπος στο θέμα αυτό. Bene. Ωραία. Τελειώσαμε. Είμαστε απόλυτα ευτυχείς κύριε Επίτροπε με τις απαντήσεις σας. Δεν ξέρω πόσοι νεοδιοριστέντες ε, επίτροποι έχουν χειροκροτηθεί όσο εσείς. Εμείς διακόπτουμε τις εργασίες μας και θυμίζω στους συντονιστές να συναντηθούν με τους βουλευτές τους, διότι στη μία θα ξεκινήσει η συνεδρίαση των συντονιστών για να αξιολογήσουμε το αποτέλεσμα αυτής της ακρόασης. Διακόπτεται λοιπόν η συνεδρίαση